Bonjour à tous. Good morning. Καλημέρα σε όλους σας, γαλλικά και αγγλικά, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Αρχίζουμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας και στα ισπανικά πλέον. Buenos días. Καλημέρα σας. Queridas y queridos. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αρχίζουμε με το σημείο 1 συνήθως έγκριση της σημερισής διάταξης. Θα πρότεινα να αναβάλουμε το 13 τι διεθνείς συμφωνίες. Είχε προβλεφθεί για αύριο το θέμα αυτό. Δηλαδή για σήμερα. Παρουσία του Αλφρέντο Πέρισου Καμπαρκάμπα, Υπουργού Εσωτερικών. Αν δεν διαφωνείτε, να αλλάξουμε. το, αύριο θα έρθουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, οι κύριοι Πέρες Ρουμπαλκάουα και Καβάνιο Ντομίγκες, αντιστοίχως, για να εκπροσωπήσουν την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου. Σημείο δεύτερο. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Αφορά την έκθεση του κυρίου Σόβερ για Σάγερ για τις ε, συμφωνίες ε, επανεισδοχής με το Πακιστάν. Στις 12 και 13 Ιουλίου θα συζητηθεί εκτός αυτή. Γιατί χρειάζεται ε, μια διαδικασία που δεν δέχεται τροπολογίες Οπότε, αν θέλετε να αντιταχθείτε σε αυτή την πρόταση, μπορείτε να την καταψηφίσετε. Τροπολογίες δεν μπορείτε να καταθέσετε. Ναι. Για το νομοθετικό ψήφισμα, 25 Ιουνίου, μέρα Παρασκευή, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία. Κυρία Φλότρο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Φλότρο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι λίγο που έχει εγγραφεί το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη τη επόμενη συνεδρίαση τον Ιούλιο. Γιατί στο Στρασβούργο, όταν συνεδριάσαμε το σκιο, με του σκιώδει και τον εισηγητή, ότι προβληματιζόμαστε για το ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να ε, εξεταστεί και να εγκριθεί αυτή η έκθεση μετά τη Λισαβόνα για πρώτη φορά σε μια χώρα που είναι κάπως ε, έτσι, ιδιαίτερη. Και εγώ είχα καταλάβει ότι θα μπορούσαμε ταυτόχρονα να έχουμε και ένα πολιτικό ψήφισμα που να διευκρινίζει τη θέση μας ως βουλευτών ως προς τη λειτουργία, τη διαπραγμάτευση, ε, αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Και εκπλήσωμαι γιατί δεν έγινε πρώτερη συνεννόηση με τους σκιώδεις ηγητές που είμαστε για να καταλήξουμε στο τι αποφασίσουμε. Καλώς κύριε Φλότρο, το σημειώνουμε. Αλλά για την ημερήσια διάταξη ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ. Κύριο Σόγκουρο, ο εισηγητή, απουσιάζει. Ε, αλλά το συζήτησα μαζί του και εγώ κατάλαβα κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε η κυρία Φλότρο. Ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε όντως αυτό το σημαντικότατο θέμα, την πρωτοβουλία και θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέλη θα έχουν πλήρη δυνατότητα να πούν ό,τι θέλουν όπως είπατε κύριε Πρόεδρε πολύ σωστά, μόνο εγκρίνουμε ή απορρίπτουμε τη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό χρειάζεται ε, πλήρη συζήτηση στην Ολομέλεια, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ δεν θα υπάρξει ψήφισμα. Μάλιστα. Συμφωνούμε για τη διαδικασία αυτή. Η κυρία Γκυγιόμ. Oui, non. Euh, πολύ γρήγορα γιατί ε, ήμουν και εγώ σε εκείνη τη συνεδρίαση με την κυρία Φλότρο και δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω ότι ε, φύγαμε από τη συνεδρίαση με αυτή τη σαφή ιδέα όλοι μας ότι πρότεινε κάτι τέτοιο εισηγητή και εμεί θα το συνοδεύαμε από δήλωση, ψήφισμα, δεν ξέρω πώ θα το πείτε και τι καθεστώ θα έχει αυτό. Ε, μια δήλωση όμω, μια ιδεκήρυξη που να έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο σχετικά με τη σύναψη αυτή τη συμφωνία και τι επόμενε που θα ακολουθήσουν. Για το πώ θα ενημερώνονται οι βουλευτέ και πώ θα έχουν τη δυνατότητα να του δίδονται απαντήσει σε ερωτήσει που επανειλημμένα έχουν κάνει. για το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας αυτής. Και επιβεβαιώνω και εγώ ότι αυτά υπόθηκαν. Τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι είχε καταλάβει και ο εισηγητής. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Το σημειώνουμε και αυτό. Ζήτω συγγνώμη, λέει ο κύριο Σάιμον Μποσουτήλ. Διαφωνώ έντονα. Είναι κανονική διαδικασία. Ε, ε, το δικαίωμα που έχει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει, να απορρίψει, ναι ή όχι, χωρίς τροπολογίες και δεν θα πρέπει να βάλουμε νέα ε, δεδομένα και να δημιουργήσουμε προηγούμενα. Θα συζητούμε και στους συντονιστές, αλλά πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με την πρόταση αυτή. be deciding at the... Θα το συζητήσουν και θα αποφασίσουν οι συντονιστές. Και προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε τη μέση διάταξη. προτείνω να ψηφίσουμε στις 12 και 13 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε στην Επιτροπή Ελευθεριών. Σημείο παριθμό 3 έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που βλέπετε εδώ, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Μαρτίου. Έχετε στους σας τα πρακτικά και αν δεν διαφωνήσετε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Προχωρούμε στο σημείο 4 Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της μετανάστευσης. Για να μας προσευχιάσει λοιπόν τα συμπεράσματα αυτά έχουμε ενώπιό μας την κυρία Άννα υφυπουργό μετανάστευσης της Ισπανικής Κυβέρνησης, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη γνωρίζετε πολύ καλά την Ανατερών. Θα θυμάστε ότι επί σειρά ετών ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της και της δίνουμε το λόγο για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της Προεδρίας και του Συμβουλίου για τη Μετανάστευση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως, το έχω συνηθίσει, αλλά να είμαι περισσότερο από την άλλη πλευρά, κάτω στο ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά το να βρίσκομαι εδώ για να επικοινωνήσουμε όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ισπανικής Προεδρίας, οπότε και θα πρέπει να προβούμε σε μια αξιολόγηση των όσων έγιναν σε σχέση με τις ε, ανακοινώσεις ε, που έγιναν από τον κύριο Κορμπάτσο στις 26 Ιανουαρίου ενεστώτος τους και θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο αφορά την μέσα διάταξη της Προεδρίας να σας πω τα θέματα τα δικά μου ως ε, αρμόδια στην κυβέρνηση για τα θέματα μετανάστευσης και θα επικεντρώσω την ενδιαφέρον μας στα εξής τέσσερα. Την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, δεύτερον για τις πολιτικές μετανάστευσης, αυτές που ασκήσαμε κατά την Προεδρία, κατά το εξάμεινο, επίσης το πρόγραμμα δράσης για τους ανήλικους, τους μη συνοδευόμενους και τα συμπεράσματα στο οποίο καταλήξαμε κατόπιν του έργου που επιτελέσαμε και τα όσα αναδεχθήκαμε, κληροδίσαμε, μας κληροδότησαν τόσο πάντων οι άλλες ε, προεδρίες. Σχέση με την αναδοχή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μεταναστών. Και όπως τα γνωρίζετε, πολύ καλύτερα από εμένα, το ότι και εσείς παρακολουθήσατε τι έγινε. Ε, ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας με κάποιες θεσμικές δυσκολίες. Τις δυσκολίες που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Οπότε και κατά κάποιο τρόπο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση για την συνθήκη και τις αντίστοιχες προσαρμογές. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας με νέους προσανατολισμού σε συνεργασία με την Κομισιόν. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαμε να ξεκινήσουμε με ένα ορθολογικό τρόπο όπως, όπως θα θέλαμε. Και αυτό πάντως το καταφέραμε λίγο πιο αργά και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε άλλο για να μην κάνουμε τίποτα, αλλά πάντως θα πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτή η δυσκολία. Τώρα, να σας πω τι έγινε με αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο αποσκοπεί να καταστεί μια ετήσια αναφορά και έκθεση σε σχέση με τα πεπραγμένα κατά το προηγούμενο έτος. Και να αναφέρονται οι προτεραιότητες για κάθε φορά το επόμενο δωδεκάμινο πρώτη ανάλυση και αξιολόγηση. Καταρχήν είμαστε ικανοποιημένοι για τα όσα μπορέσαμε να προωθήσουμε. Πρώτα-πρώτα, αυτό το σύμφωνο βασίζεται σε κάποιες δεσμεύσεις, κάποιες αρχές. Αυτά όλα ήταν το αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης που πάντα καθορίζει είπαμε τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο όπως σας προανέφερα έχουμε αυτή την αξιολόγηση, αξιολόγηση του συμφώνου ούτως ώστε να δούμε, επί τη βάση των όσων συμφωνήσαμε, να δούμε τι θα γίνει με την πολιτική μετανάστευση. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιους μηχανισμούς συντονισμούς. Και επίσης τη χρήση κάποιων δικτών όπως και στην αλυσίδα της Αραγώσας καθορίστηκε, αλλά επίσης να, δούμε τι γίνεται με τη Frontex που ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο πολιτικής. Ε, και στη χώρα μας αυτά τα αντιμετωπίσαμε και είδαμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το ότι είχαμε κάποια συρρήγνωση των, ε, της εισόδου λαθρομεταναστών. Βέβαια αυτό δεν αφορεί μόνο τη χώρα μας, αφορά το σύνολο των ενωσιακών σύνορων επίσης και για το άσυλο, να δούμε τι έγινε, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει, μια που θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους στόχους της πολιτικής μετανάστευσης και όλα αυτά στο πλαίσιο του διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι πετύχαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία στο Συμβούλιο γιατί γνωρίζετε ότι στο Συμβούλιο καθένα έχει τι δικέ του ευαισθησίε. Οπότε και αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή αυτή η αξιολόγηση του συμφώνου, θα ωφελήσει και θα εξυπηρετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο διακρίνεται από διαφάνεια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει εποπτεία του τι γίνεται στο Συμβούλιο, θα γίνεται μια αξιολόγηση, απολογισμός των πεπραγμένων, και ταυτόχρονα θα βοηθάει στην, στον προγραμματισμό για την ε, επόμενη κάθε φορά περίοδο. Άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι το πρόγραμμα της πολιτικής μετανάστευσης. Της νόμιμης μετανάστευσης. Έτσι τη λέμε. Νόμιμη μετανάστευση. Αλλά βέβαια αυτό και για μένα είναι ε, κάπως πλεονασμό γιατί αφού λέμε για πολιτική μετανάστευση εννοούμε την νόμιμη μετανάστευση. Αλλιώ μιλούμε για παρανομία. Και επομένω, αυτό το πρόγραμμα που αφορά την μετανάστευση αποτελεί μία προτεραιότητά μας. Και δεν μπορέσαμε, όπω γνωρίζετε, να κάνουμε τίποτα όσον αφορά αυτούς τους εποχιακού εργαζομένου και όσον αφορά την μεταφορά από τον ένα κλάδο στον άλλο κάποιων εργαζομένων, γιατί η κατάσταση ε, θεσμικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, οπότε και η Κομισιόν δεν μπόρεσε, δεν βρήκε το χρόνο για να παρουσιάσει κάποιες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Και είχαμε κάποιες ε, επαφές, διαπραγματεύσεις όσον αφορά την μία ενιαία άδεια. Αυτά όλα τα συζητήσαμε, τα προσιάσαμε στο Συμβούλιο όσον αφορά ένα πεδίο εφαρμογή ευρύ. Ούτω ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο αναφορά όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων. Θεωρώ ότι έγιναν βήματα πρόοδου σημαντικά. Μπορέσαμε επίσης να περιλάβουμε τις δικές σας προτάσεις και της ε, ε, Επιτροπής ε, Κοινωνικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου και για τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ γιατί πρόκειται για μια συνεργασία που είχαμε μαζί σας που έγινε με αμοιβή εμπιστοσύνη, έγινε με διαφάνεια, έγινε με τρόπο επαγγελματικό. Οπότε έτσι και βάλαμε τις βάσεις για να προχωρήσουμε άμεσα. Τώρα προκειμένου να ε, συνεργαστούμε με τη Βελική Προεδρία και έτσι αυτή η οδηγία για την ενιαία άδεια να ε, υλοποιηθεί. Αλλά πάντως βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στην Βελική Προεδρία και θα γίνει η διεκπαιρέωση του το επόμενο εξάμεινο. Υπάρχει τώρα και ένα άλλο θέμα το οποίο για την Ισπανική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για το πρόγραμμα δράση που αφορά τους μη συνοδευομένους ανηλίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοούμε για κάποιου που έρχονται με δύο διαφορετικές ροέ. Ε, ροές. Γιατί είναι πρώτα-πρώτα η ροή των προσώπων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναζητήσουν καταφύγιο και άσυλο και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιες άλλες ροές. Εκείνους δηλαδή οι οποίοι σκοπεύουν να αναζητήσουν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ανήλικοι, πολλές φορές είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά που θεωρούν ότι μπορούν να αναζητήσουν την, την ευκαιρία εδώ στην ε, Ένωση και προσκρούν σε κάποια πρακτικά ή άλλα προβλήματα. Οπότε θέλαμε να, δούμε κάτι, να, τι μπορεί να γίνει ως προς αυτό με κάποιο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα έχει ως θεμέλιο μια βασική ξεκάθαρη αρχή που θέλω να σας τονίσω. Ότι δηλαδή θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε να θεωρούμε ότι κυρίαρχο συμφέρον είναι αυτό του ανηλίκου. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έχουμε αυτό το πρόγραμμα που προβλέπει τρεις διαφορετικές δράσεις που θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτα πρώτα η πρόληψη της μετανάστευσης υπό συνθήκες που καθιστούν πάρα πολύ ευάλωτα αυτά τα άτομα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε το να θέλει κάποιος να είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο να υφίστανται αυτά τα άτομα ε, να υφίστανται πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, δηλαδή να είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Επίσης ε, έτσι, θέλουμε μέσα αυτό το πρόγραμμα να, να δούμε πώς θα τους υποδεχόμαστε και πώς θα τους προστατεύουμε αυτούς τους ανηλίκους. Επίσης προβλέπονται κάποιες διατάξεις συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Τέλος, προς το συμφέρον των ανηλίκων όπου είναι δυνατόν ε, να υπάρχει συνένωση ή επανένωση της ε, οικογένειας και να είναι δυνατόν να υπάρχει ασφαλής επιστροφή. Επίση, θέλω να σα τονίσω ότι όλοι αυτοί οι δέσμοι των μέτρων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτή τη δράση σε σχέση με του μη συνοδευμένου ανηλίκου, όλα αυτά λέω είναι περιπτωσιολογική ρύθμιση. Δεν υπάρχει μια προηγουμένω ληφθή απόφαση για αυτό το πρόγραμμα δράση σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά αυτού του ανηλίκου. Απλώ προβλέπεται ανάλυση αναπερίπτωση. Σε σχέση με την κάθε περίπτωση λοιπόν και επί τη βάση της οποίας αποφασίζεται το τι λύση θα δοθεί σε κάθε περιστατικό. Και πάντοτε βασί το πώς θα ωφεληθεί αυτό το παιδί. Άλλες επιτυχίες, αν μου επιτρέπετε να σας πω, που μας κάνουν περήφανος, είναι τα συμπεράσματα της υπουργικής διάσκεψης της Σαραγώσα όσον αφορά την ένταξη. Πήραμε τη σκητάλη από άλλε σε αυτό το θέμα, πήραμε τη σκητάλη από άλλε διασκέψει αντίστοιχε και σα ε, τονίζω ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε το επιτελεστέν έργο των Υπουργών για το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό για μας. Η ΔΕ Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών εκπροσωπήθηκε μέσω του Προέδρου της. Αυτό μας χαροποιήσει πάρα πολύ γιατί θεωρούμε ότι Πρέπει να συνεργαστούμε με την ε, Επιτροπή σας και Γύρω με το Κοινοβούλιο. Τώρα, τα βασικότερα θέματα εδώ είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση με τη στρατηγική για το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση με τους μετανάστες. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες δράσεις ε, κατάρτισης γιατί πρόκειται για ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο ανθρώπινο, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο να κινηθεί σε αυτό το τοπίο του 21ου αιώνα, το τοπίο της παγκοσμιοποίησης. Οπότε είπαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη γραμμή πλεύσης σε συνέπεια με τη στρατηγική μας για το 2020 και με το σύνολο των προβλεπωμένων μέτρων. Δεύτερον, κάτι το οποίο και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί το Κοινοβούλιο, απασχολεί την Επιτροπή σας, το πώς θα μπορούσαμε να παρεύουμε σε κάποιες γειτονίε, σε κάποιες ζώνες με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού μεταναστών. Όπου δηλαδή το θέμα δεν είναι την μετανάστευση, είναι το ότι εκεί σοβεί φτώχεια και άλλα προβλήματα και ότι υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να δούμε το πώς θα γίνει ούτως ώστε αυτοί να έχουν το αίσθημα του, του ανήκειν, το αίσθημα του συμμετέχειν σε, σε, σε κάποιες καταστάσεις ε, κοινωνικά δύσκολες περίπλοκες. Τώρα κάτι άλλο το οποίο από πλευρά πολιτική είναι λιγότερο σεξ, λιγότερο ελκυστικό, αλλά νομίζω ότι για τη δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πώς θα κάτσουμε να επεξεργαστούμε κάποιους ε, δείκτες, τόσο ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε, να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα προγράμματα αυτά και να μπορούμε να έχουμε και συγκρισιμότητα όσον αφορά κάποιες πρακτικές που ισχύουν στις διάφορες χώρες μας. Έχουμε και σχετική συνέντευξη τύπου. Πάση τόσο, αυτό μας απασχόλησε πάρα πολύ και το ζητήσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσει κάποιο είδους πιλωτικό πρόγραμμα αυτό το στόχο. Στόχο του να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις πολιτικές ένταξης και να υπάρχει συγκρισιμότητα. Προτεραιότητες και στόχοι που σας είχαμε τότε αναπτύξει εδώ, το έκανε η Προεδρία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας. Αυτές οι προτάσεις, οι αναγγελίες νομίζουμε ότι ολοκληρώθηκαν. Τώρα παίρνει τη σκητάλη Βελική Προεδρία. Ευχαριστώ να απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσει, αλλά και με χαρά μα να δούμε κάποιε δικέ σα προτάσει που θα τι επεξεργαστούμε στο μέλλον στα πλαίσια τη τροϊκα. Ευχαριστώ. Την κυρία Τερών και όπως είπαμε προηγουμένως ακολουθεί η ανταλλαγή απόψεων. Για όλα τα μέλη που θέλουν το λόγο μπορούν να το ζητήσουν τώρα. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ, ορίστε. Κύριε Δίας Δεμέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Υφυπουργό για την παρουσίασή της για τα τέσσερα σημεία ε, τα οποία κάλυψε. Σύντομα, έχω κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω τις οποίες μου έχετε ενδύσει όμως, καλύφθηκα από τα τέσσερα σημεία στα οποία αναφερθήκατε. Ε, του συμφώνου, ε, του συμφώνου ασύλου και μετανάστευσης, συγγνώμη. Η πολιτική μετανάστευση, η μη συνοδευμένη ανήλικη και τα θέματα της ε, Θα ήθελα λοιπόν σύντομα να σας ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις. Για παράδειγμα, σχετικά με το πρώτο. Η ασυνόδευτη ανήλικη. Είναι πολύ σημαντική και πολύ αναγκαία η πρότασή σας. Αλλά πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων. Πού βρίσκεται η πρόταση αυτή. Σε ποιο στάδιο. Ερώτηση δεύτερη. Τονίσατε την υποστήριξη ε, της οδηγίας που είναι γνωστή εδώ ως οδηγία Θέρκας και ότι ανεπιφύλακτα υποστηρίζεται την οδηγία αυτή. Πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων σήμερα. Είναι η ίδια ερώτηση που σας έκανα για το προηγούμενο θέμα. Διαδικαστικά, πολιτικά, σε ποια φάση βρίσκεται. Τρίτον, γιατί Frontex. Γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός αυτός, Frontex, είναι ουσιαστικά συντονισμός των μέσων που τίθεται στην υπηρεσία των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν κάποιες οξύες καταστάσεις και κρίσεις. Δεν είναι υποκατάσταση των δικών τους ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Ποιο είναι το προφίλ του νέου οργανισμού Frontex με ορίζοντα έτσι χρονικό το 2013. Ποιες θα είναι όμως οι νέες εξουσίες και αρμοδιότητες. Κατά την άποψη την κρίση της Ισπανικής Προεδρίας οφείλει να έχει ο Frontex και δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή. Και τέλος ήθελα να σας κάνω ένα σχόλιο, μάλλον ε, θεωρητικό, φιλοσοφικό. Χαίρομαι πολύ που ο πρόεδρος πήγε στη διάσκεψη των πρόεδρων στη ε, Σαραγώσα για να μιλήσει για την ενσωμάτωση. Αλλά αυτό είναι εθνική, ξέρετε, αρμοδιότητα, δεν είναι κοινοτική. Καλό είναι να συζητούμε κάποιες πρακτικές και ε, πολιτικές, αλλά στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αλληλέγγυοι. Και κατά την άποψή μου η αλληλεγγύη για την ενσωμάτωση περνάει και ε, μετράται από τέσσερις ε, παραμέτρους που δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν και αυτά ονομάζονται εργασία, σχολείο, υγεία, στέγη. Πολύ ωραίο είναι λοιπόν να κάνει κανείς δηλώσεις προθέσεων. Ακόμα ωραιότερο και καλύτερο να συντονίζουμε και να συγκρίνουμε καλές πρακτικές. Αλλά ουσιαστικά η ενσωμάτωση των μεταναστών είναι εθνική αρμοδιότητα και όχι κοινότική. Αυτό άλλωστε υπόθηκε κιόλας και συμφωνώ και στο Κοινοβούλιο από πλευρά Ισπανική Προεδρία. Η ίδια Ισπανική Προεδρία το δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτό συνιστά εθνική και όχι κοινοτική αρμοδιότητα. Ποια θα πρέπει να είναι όμω η αλληλεγγύη μα για να καταφέρουμε αυτά τα σημαντικά και επαναλαμβάνω ποια είναι. Τέσσερα κατά την άποψή μου. Η εργασία, το σχολείο, η υγεία και η στέγη. Ε, Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου για την εργασία σας και την παρουσία σας και εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος σας ζητούσα ε, μερικές διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, ο κύριος Μωράης. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω την κυρία Τερών Έμαθα πολλά από την Άννα. Ξέρω ότι έχει πάει από την άλλη πλευρά, ε, από τα έδρανά μας. Ε, στο Κοινοβούλιο εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με την ορολογία και με τον όρο της μετανάστευσης. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Νομίζω ότι κάλυψατε πάρα πολλά ζητήματα για τη μετανάστευση. Πήγατε μέχρι και το άσυλο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ευρύτερη άποψή σα για δύο-τρία θέματα. Αναφέρατε πολλά, εγώ επέλεξα μερικά που είναι σημαντικά για την ομάδα μας. Είπατε ότι τα δικαιώματα των μεταναστών είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά και για την αγορά εργασίας. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε εμείς από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας και θα θέλαμε να ξέρουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι θέμα διαφωνίας μεταξύ των δύο επιτροπών. Αυτό μας ε, απασχολεί πάρα πολύ και θα θέλαμε να ξέρουμε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ε, ε, καλύψατε με την προηγούμενη απάντη, με την, καλύψατε με τα σχόλιά σας τη δεύτερη ερώτησή μου. Αλλά ως υπουργό που έρχεστε τώρα προς το τέλος της προεδρίας, ποια είναι η άποψή σας για το πακέτο του ασύλου. Γιατί οι συζητήσεις που έχουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θίγουν τον πυρήνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και το Συμβούλιο στο θέμα του ασύλου. Είμαστε σε μια θέση αυτή τη στιγμή όπου πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα και να ακολουθήσουμε τις σωστές διαδικασίες. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο στο Συμβούλιο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Για μας το Κοινοβούλιο θέλουμε να διατηρήσουμε το πακέτο όσο το δυνατόν περισσότερο στην ακαιρεότητά του, αλλά κατανοούμε ότι στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να μην συμβεί. Ε, θα θέλαμε να δούμε αυστηρές προθεσμίες, σαφείς στόχους και μια καλύτερη υποδοχή από πλευράς Συμβουλίου για την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να πάρουμε. Δεν θέλουμε να ταλματώσουμε. Ποια είναι λοιπόν η γενική σας άποψη γι' αυτό. Και τέλος για το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι ο αγώνας που δώσαμε για την κοινωνική ένταξη και που ανάγεται πίσω την εποχή που ήσασταν κι εσείς εδώ η κοινωνική ένταξη είναι κάτι που αντιμετωπίζεται καλύτερα σε τοπικό επίπεδο, όπως ξέρετε πολύ καλά, και μερικές φορές σε εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ρητή νομική βάση για την κοινωνική ένταξη. Αυτή είναι η αλλαγή. Και αφού έχουμε αυτή τη νομική βάση, θα ήταν καλό να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας τώρα εδώ στο τέλος της Προεδρίας είναι πραγματικά εφικτό να σημειωθεί πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ένταξη με βάση τις κοινέ βασικές αρχές. Ξέρω ότι δεν αναφέρεται η ένταξη πια πολύ στο Κοινοβούλιο, δεν γίνεται και πολλής λόγος ε, γι' αυτό. υπάρχουν κάποια πολύ καλά μέτρα που έχουν ήδη αναλυφθεί, όπως η νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Αυτά έχουν επιτευχθεί. Ποια είναι τώρα η άποψή σας που θα δώσετε τη σκητάλη στην Βελγική Προεδρία. Ε, τι, ποιο είναι η κληρονομιά που μας έχει μείνει στα χέρια μας για την κοινωνική ένταξη. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριος Μπουζούτιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ε, το καλωσόρισμά μου ε, προς την Υπουργό, ε, να την ευχαριστήσω για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι αν δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της μετανάστευσης στο πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, θα πούμε ότι δεν έγιναν και πολλά, <laughs> δεν έχουμε και πολλά Νομίζω όμω ότι η Ισπανική Προεδρία μπορεί να συγχωρηθεί για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι ότι περάσατε ένα δύσκολο εξάμεινο. Ε, δεν υπήρχε επίτροπο όταν ξεκινήσαμε και δεν υπήρχε και πλάνο εργασία για την επόμενη θητεία της Επιτροπής. Το δεύτερο είναι ότι είχατε ένα σχέδιο δράση που, παρουσιάσατε ένα σχέδιο δράση που συνδέεται με τη Στοκχόλμη και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό αυτό. Κατα με βάση αυτό το σχέδιο δράσης ξέρουμε προς τα που θα πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια και έχουμε και ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για το σχέδιο δράσης, γιατί αυτό έχει κρίσιμη σημασία για τις εργασίες της Επιτροπής μας, αλλά και γιατί δίνεται το σωστό μήνυμα ότι τα δικαιώματα των πολιτών είναι εξίσου σεβαστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Για το πακέτο του ασύλου, ο Κλόντ έκανε τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω κι εγώ, άρα δεν θα πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Ε, για τη μετανάστευση θα ήθελα να πω το εξή: Είναι σωστό να υπάρχει μια ισορροπημένη πολιτική μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης ε, μετανάστευσης. Η ομάδα μας, το ΕΛΚ, είναι πλήρως διατεθειμένο να συμμετέχει σε επικοδομητικό διάλογο για να εκπονήσουμε νέα εργαλεία στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό δεν θα είναι αξιόπιστο αν δεν συνοδευτεί από μια αυστηρή πολιτική κατά της ε, λαθρομετανάστευσης. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Εάν πρόκειται να εκπονήσουμε εργαλεία για τον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, πρέπει να εκπονήσουμε εργαλεία και για τον τομέα της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί αν πρόκειται να ανοίξουμε μια νόμιμη οδό εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει ταυτόχρονα να κλείσουμε όλες τις παράνομες εισόδους από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν βρίσκονται. Και αυτά πρέπει να τα επιδιώξουμε με σταθερές πολιτικές μέσω του οργανισμού Frontex αλλά και μέσω των συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε διαρκώς να υπονομεύουμε, να υποσκάπτουμε ή να αγνοούμε τη σημασία των συμφωνιών επανεισδοχής που αφορούν άτομα που παράνομα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για άτομα που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων ε, στους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική μας για το άσυλο. Οι παράνομοι μετανάστες όμως, οι λάθρο μετανάστες, ε, πρέπει να γίνουν δέκτες ε, του κράτους δικαίου. Να εφαρμοστεί σε αυτούς το κράτος δικαίου. Έτσι το βλέπω εγώ. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η άποψη της Ισπανικής Προεδρίας τώρα που πλησιάζει στο τέλος της εξάμηνης προεδρίας της και συγκεκριμένα για τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της νόμιμης μετανάστευσης και της λαθρομετανάστευσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε και πάλι κυρία Τερών. Ε, μερικές από τις ερωτήσεις που είχα να σας κάνω έγιναν. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ακούσουμε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τη μετανάστευση, με την ένταξη των μεταναστών και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι γεγονός βεβαίως ότι θα πρέπει να είμαστε θεραλέοι ε, στις συζητήσεις μας και να μην έχουμε ψευδο Έχω την εξή ερώτηση. Όλο και περισσότερο βλέπουμε σήμερα και ακούμε φωνές που χρησιμοποιούν τη μετανάστευση για να στιγματίζουν κάποιους ανθρώπους και θα μπορούσαμε να πέσουμε στον πειρασμό να αναζητούμε μέτρα που όλο και περισσότερο καταδικάζουν παρά βοηθούν εκείνους που θέλουμε να βοηθήσουμε. Και θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να σας μιλήσω για μια πολύ ειδική περίπτωση. Είναι ε, το Ισλαμικό φουλάρι και η μπουρκα σε διάφορα κράτη και πώς χρησιμοποιείται. Δεν είναι γενικευμένο σε όλη την Ευρώπη με το ίδιο τρόπο. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ε, ανάλογα με τις περιπτώσεις και ανάλογα με τις χώρες. Σε άλλες χώρες υπάρχουν περισσότερες και σε άλλες λιγότερες. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ε, πολιτιστικού σχετικισμού για να υπερασπιστώ το ε, απαράδεκτο. Απλώς θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα κάθε φορά. Και θέλω να σας κάνω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό το θέμα που είναι επιτάπητος και αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, αριθμητικά ενώ δεν είναι πρόβλημα πια σε κάποια μέρη της Ευρώπης και μιλώ για την Καταλωνία αλλά ε, ε, η συζήτηση έχει αρχίσει και νομίζω ότι μέχρι ενό σημείου είναι τεχνητή συζήτηση διότι θέτει ένα πρόβλημα που δεν είναι από μόνο του πρόβλημα Αντίθετα, ορισμένα από τα μέτρα που ορισμένοι προτείνουν, όπως η πλήρη ε, απαγόρευση να κυκλοφορούν σε δημοσίους χώρους ή να προσφέρουν σε δημοσίους ε, χώρους γυναίκες που φορούν Ισλαμική μαντήλα ή ε, μπουρκα, μπορεί να οδηγήσει σε διπλή διάκριση βάρους τους δεν λέω ότι δεν πρέπει να το συζητούμε, λέω ότι ε, κατεύθυνση παίρνει η συζήτηση, γιατί καμιά φορά ε, μα κατηγορούν για σχετικισμό. Καθόλου, καθόλου. Να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά με τρόπο έτσι ε, σόφρονα και συνεπή. Και έχω την εξή άμεση ερώτηση. Στο βαθμό που ακόμα μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα προληπτικά και όχι κατασταλτικά, ποια είναι τα μέτρα που σκέφτεστε, που μελετάτε, που θα μπορούσατε να εξετάσετε ακριβώς για να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο ανθρώπινα. Και η πίεση να μην είναι στους ώμους της γυναίκας που είναι θύμα, αλλά εκείνου που την υποχρεώνει να ζει σε αυτή την κατάσταση. Και πολύ συγκεκριμένα, πολλές φορές είναι οι ίδιοι οι μάμιδες. Ευχαριστώ, κυρία Λάμπερτ. Ε, thank you. And, um... Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θα ήθελα να κάνω μια-δυο ερωτήσεις που συνδέονται με την ε, συζήτηση για την ε, ενιαία άδεια. Ε, πολλοί αρχίζουν να ρωτούν ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ενιαίας, ε, της μίας και μόνης άδειας στο πλαίσιο της κοινή μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μερικοί από εμά βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ζητούν για πολύ μεγάλη ευελιξία για το εργαλείο αυτό. Εσείς θέλετε να δώσετε τον ίδιο τίτλο σε αυτό το εργαλείο. Ε, τι θα προσφέρει στην κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μετανάστευση και σε σχέση με αυτό, όπως είπαμε ήδη, ε, τώρα το αντιμετωπίζουμε το θέμα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με την Επιτροπή Απασχόλησης και αυτό νομίζω εγείρει ένα ερώτημα για το κατά πόσο οι ανησυχίες και οι παράμετροι της απασχόλησης και, και της κοινωνικής συζήτησης, η αγορά εργασίας, η δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσο όλες αυτές οι παράμετροι και οι ανησυχίες ε, μεταφυτεύονται ε, στον τομέα της μεταναστευτικής ε, πολιτικής. Υπάρχουν κάποια πολύ θετικά επιχειρήματα που ακούγονται από την πλευρά της μετανάστευσης, αλλά η πλευρά των εσωτερικών υποθέσεων, αν θέλετε, ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς να κρατήσουμε τους περισσότερους έξω και να βρεθεί η σωστή νομική βάση για να κρατήσουμε κάποιους ελάχιστους μέσα. Ε, δηλαδή τελικά ποια είναι η συνεργασία, πώς συνεργάζονται οι Υπουργοί Απασχόλησης και οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων σε αυτό το υψηλό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί αυτή η κοινή προσέγγιση που συζητούμε εδώ. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Μια πολύ απλή ερώτηση έχω να κάνω. Ε, πάει πάνω από ένας χρόνος που υιοθετήθηκε η μπλε κάρτα. Θα ήθελα να ξέρω τι πρόοδος έχει σημειωθεί στα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής. Ε, πώς έχουν οι εξελίξεις, έχει εφαρμοστεί και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα, πώς οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει την μπλε κάρτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδίως την Υπουργό, ιδιαίτερα την Υπουργό για την ε, παρουσίαση των εργασιών ε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Εκτίμησα όλος ιδιαίτερος ε, ορισμένους από τις προβληματισμούς της, ορισμένους από τους στόχους που υπογράμμισε εκ νέου ο Υπουργός σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα ή μάλλον κυρίως την ανάγκη ενίσχυσης της εμπειρίας της Frontex. Προφανώς είναι μια εμπειρία εξόχως ε, ευρωπαϊκή και υπάρχει και ο στόχος ε, να προχωρήσουμε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ε, ακριβώς γιατί Ακριβώς επειδή συμφωνώ και πιστεύω ότι εκφράζω και την άποψη όλων, πιστεύω ότι συμφωνούμε με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην μετανάστευση. Θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για μια μετανάστευση με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπουζούτιλ. πράγματι πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των νόμιμων μεταναυστών και να υπάρχει σωστή υποδοχή τους και σωστή κοινωνική ένταξη, αλληλεγγύη και υποδοχή όπως είπα, αλλά απαιτούνται και κανόνες πολύ αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Με μεγάλη μου όμως ευχαρίστηση άκουσα κάτι που εσείς ως υπουργός υπογραμμίσατε και συγκεκριμένα την ένταση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων. Είναι πάρα πολλοί οι ανήλικοι που βρίσκονται σε, αυτές τις, σε αυτή την επισφαλή κατάσταση και δεν πρέπει ως Ευρωπαίοι να επιτρέψουμε την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερα τροτής κατηγορίας ε, δεν, μπορούμε, δεν μπορούν να τυχαίνουν της ίδιας μεταχείρισης οι ανήλικοι όπως οι ενήλικοι. Και γι' αυτό στην νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει σε λίγο, με την οποία θα ασχοληθεί σε λίγο η συγκεκριμένη Επιτροπή του Κοινοβουλίου μας, αφορά ακριβώς τους ασυνόδευτους ανήλικους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπρόνζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έγινε καμιά μελέτη για τα προβλήματα που υποδέχονται μετανάστες ε, ανειδίκευτους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των ε, ε, εργαζομένων στην υγεία. Βρετανική πολιτική έχει προάγει πάρα πολύ το εθνικό σύστημα υγεία της και το έχει κάνει ελκυστικό ε, για τους ε, ξένους εργαζόμενους. Ε, προσελκύονται πάρα πολύ από όλο τον κόσμο και πολλές δαπάνες γίνονται για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εμπειρία τους για να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους λαούς. Θα έπρεπε πιστεύω οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν πίσω στις πατρίδες τους και να χρησιμοποιούν την κατάρτιση και την εμπειρία τους και αντί να ληστεύεται ο τρίτος κόσμος από το νοσηλευτικό του και το ιατρικό του προσωπικό. Έρχομαι τώρα στον πόλεμο του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε ένα μελλοντικό ε, πόλεμο κατά του Ιράν για να αποφύγουμε ένα νέο κύμα ετούντων ασύλου όπως συνέβη με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Άκουσα τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται ως ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά ως ε, ε αναλώσιμα της παραγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταβάνης. Έχω μια ερώτηση, θα σας την πω κυρία Υπουργέ, ή στα πορτογαλικά. Falamos acerca ε, γίνεται λόγος για τη μετανάστευση, την νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών. Εδώ στο Κοινοβούλιο δεν είναι ενιαία η άποψη όλων των πολιτικών ομάδων για αυτό το θέμα. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πολιτική για αυτό το θέμα ε, είναι φυσικό να είναι πολλές οι απόψεις και πολλές οι πολιτικές. Έτσι δεν είναι άλλος ε, ακολουθεί πιο ανοιχτή πολιτική, άλλος πιο κλειστή, πιο φιλελεύθερη, πιο κατασταλτική. Εγώ προτείνω μια γραμμή πιο φιλελεύθερη, πιο ανοιχτή και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το υπερασπιστώ. Έχω την αίσθηση ότι στην Ευρώπη ε, μέγα τμήμα της κοινωνίας των πολιτών προτιμάει μια πιο κλειστή γραμμή και πιο κατασταλτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. που βεβαίως πάντα αυτό υπερισχύει στον πληθυσμό. Γιατί το λέω αυτό. Όπως και οι περισσότεροι παρόντες, αν όχι όλοι, ε, θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσεις τη λαθρομετανάστευση είναι να έχεις μια σωστή πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση. Το είπε και η κυρία Υπουργό άλλωστε. Και είναι προφανές και αυτονόητο ότι δεν θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε προς την ε, καταστολή και μόνο, να πατάξουμε τη λαθρομετανάστευση. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε μία διέξοδο στην νόμιμη μετανάστευση, από νομίμους διάβλους. Και σε ό,τι αφορά τώρα την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Σε δύο σημεία συμφωνώ με τον αγαπητό φίλο και Δίας Ντεμέρα. Παρόλο που η πολιτική κοινωνική ενσωμάτωση είναι εθνική αρμοδιότητα και όχι κοινωνική, κοινοτική, συγγνώμη, έχουμε και κοινοτικέ προσεγγίσεις, ας πούμε, για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά για τη δημοκρατία. Και θα ήθελα να θυμίσω και πάλι αυτό που είπε ο κύριο Δία μέρα. Δεν είναι μόνο η εργασία, το σχολείο, η υγεία και η στέγη, αλλά και η συμμετοχή στην κοινωνία των μεταναστών. Και έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό και τα θεσμικά της όργανα. Ακόμα και με προτάσεις, νέες ιδέες για τη μετανάστευση και μία από αυτές ε, που έχει ήδη ακουστεί είναι το δικαίωμα του εκλέγην και ε, της απόκτησης της ε, ηθαγένειας για τους μετανάστες ακόμα και αν βρίσκεται στο τέλος της, η Ισπανική Προεδρία μπορεί να δώσει ένα θετικό μήνυμα. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι μετανάστες είναι στην πρώτη γραμμή της ίδιας τους της ενσωμάτωσης όταν συμμετέχουν στην κοινωνία. Και πώς ε, ήδη συμμετέχουν, πληρώνουν φόρους, ε, εργάζονται, άρα θα μπορούσαν να ψηφίζουν και στις εκλογές. Τώρα έχω και μία πρόταση και μία συγκεκριμένη ερώτηση για τους πρόσφυγες. οι πρόσφυγες είναι πολύ σημαντική συνδετική κρίκη της κοινωνίας με τους μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει πολλά πράγματα. Θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προοπτικές που βλέπετε. στο Κοινοβούλιο έχουν γίνει εκθέσεις, δύο μάλιστα. Το Συμβούλιο τι λέει σχετικά για τους πρόσφυγες και τι θέλει ακόμα να κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί η Προεδρία της, η Ισπανική Κυβέρνηση και πώς θα διευκολύνεται τη μετάβαση προς τη Βελγική Προεδρία. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία μονάδα επανεγκατάστασης ε, των ε, προσφύγων επαναπροώθησης ε, υπάρχουν χρήματα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό και δεν μπορούμε να παρεμποδίζουμε τις εξελίξεις λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και διοικητικών και διαδικασίες που θα μπορούσαν να, κρατούν δύο εβδομάδες, κρατούν δύο χρόνια ολόκληρα, με προβλήματα για οικογένειες, παιδιά των προσφύγων. Όλοι συμφωνούμε από το ΠΕΠΕ, από το ΕΛΚ μέχρι την ΚΟΕ για αυτό το θέμα. Υπάρχει και ένα σχέδιο πιλωτικό για σύνδεση των Δήμων και κοινοτήτων με τους πρόσφυγες ε, και τους μετανάστες για να αντιμετωπίσουμε τα νέα κύματα έτσι ώστε ε, να είναι ακριβώς ένα σύνδεσμος οι πιο παλιοί και εγκατεστημένοι εδώ μετανάστες και πρόσφυγες με τους νέους που έρχονται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω γι' αυτό, να σας επιστήσω την προσοχή επίσης στη δυνατότητα ενίσχυσης αυτού του προγράμματος στη χώρα σας υπάρχουν δήμοι και κοινότητες που κάνουν αυτά τα προγράμματα επαναγκατάστασης των προσφύγων. Ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος από τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε με πολύ ακριβή και περιστατωμένο τρόπο αναφερθήκατε στην επόμενη πρόταση για την οδηγία για την εποχιακή εργασία, για την εποχιακή απασχόληση. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα και ανταποκρίνεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Ε, μιλώ για το προφίλ εργασίας. Είναι μία μη αξιοπρεπής εργασία, μία φτωχή εργασία. Και ακριβώς το ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω είναι το εξής. Η φιλοσοφία αυτού του νομοθετήματος λαμβάνει υπόψη τις προσανατολισμούς που εκπώνησε η δική σας κυβέρνηση η άδεια παραμονής των επαρχιακών εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες τους δίνει πραγματικά ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργεί πραγματικά ευκαιρίες απασχόλησης. Ευχαριστώ κύριο Κίρχοπ. Ευχαριστώ πρόεδρε και να με συμπαθά κύριε Υπουργό που δεν ήμουν εδώ να ακούσω την εισήγησή της αλλά ε, αυτό που θα σας πω εάν τυχόν το έχει θίξει κάποιος άλλος δεν χρειάζεται να το πω. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι όχι τόσο ο τρόπος διαχείρισης των μεταναστών ε, και εκείνων που έχουν θύματα δουλεμπορίου για να μπουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλω να πω κυρίως κάτι το οποίο αφορά τη σχέση με τις τρίτες χώρες που σε πολλές περιπτώσεις ευθύνονται για αυτές τις ροές του πληθυσμού. Και ε, α, συγκεκριμένα Δυτική Αφρική, Βόρειος Αφρική, Για να δούμε, υπάρχει και κάποιο είδου δυναμική ενέργεια που έχει αναλάβει η Προεδρία όσον αφορά αυτέ τι χώρε, ούτω ώστε να του δείξει ότι πολλέ φορέ αυτέ είναι η πηγή των ε, προβλημάτων και άρα θα πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του για τα αποτελέσματα των πράξεων. Γιατί οι δύο χώρε τη περιφέρεια ε, τη της Ένωση θα πρέπει ακόμα και με την βοήθεια τη Frontex να φέρουν δυσανάλογα το βάρο αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής. Εχθές είχαμε την κυρία Ρέντινγκ που μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και με βάση αυτό το χάρτη ελέγχει την κατάσταση και αυτός ο χάρτης, ξέρετε, δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το Κοινοβούλιο και ε, όλα τα θεσμικά όργανα. Η Ισπανική Προεδρία, τι κάνει, ε, πώς φαντάζεται το Συμβούλιο να επεξεργάζεται αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα αφορά την απελευθέρωση της θεώρησης ε, διαβατηρίων. Έγιναν μεγάλες διακηρύξεις και εξαγγελίες στο παρελθόν βαρύγδουπες για αντίστοιχη απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, με την Τουρκία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για επιχειρηματίες, για φοιτητές και επίσης η Συμφωνία Επανιζωχής. Έχετε τίποτα πιο πρόσφατες εξελίξεις υπόψη σας, έχει προχωρήσει καθόλου αυτό το θέμα, έχετε συμφωνήσει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε τώρα να απαντήσετε όλες μαζί τις ε, τεθείς σας ερωτήσεις. Κυρία Τερών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν μου επιτρέπετε να απαντήσω πρώτα πρώτα αυτό το είπε ο κύριος Ρωμέβα. Για το οποίο δεν είχε σχέση με το πρόβλημα της Προεδρίας, αλλά με μεγάλη μου χαρά να του πω την γνώμη μου όσον αφορά το θέμα. Για το τι κάνουμε στην Ισπανία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι γίνεται συζήτηση, ότι έχει αποκρισταλώσει κάποια θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις σήμερα κιόλας θα συζητηθεί στην Ισπανία ένα σχέδιο ψηφίσματος. Προέρχεται από μια πολιτική ομάδα, πολιτικό κόμμα ζητούν να απαγορεύεται να, καλύπτουν, να καλύπτονται οι γυναίκες. Οπότε, στη Γερουσία υπάρχει μια αλλακτική πρόταση από όλες τις πολιτικές τα άλλα πολιτικά κόμματα και εγώ προσυπογράφω αυτή την πρόταση, ότι δηλαδή να υπάρξει απόρριψη απόρριψη απόλυτη και κάθεται για οποιοδήποτε είδους διακριτική μεταχείριση και περιστολή του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια της γυναίκας. Δεν ε, πάση τόσο να είναι σαφές ότι τέτοιου πρακτικές και, και, και, και Ενδύματο ότι είναι απαράδεκτα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς ταυτόχρονα όμω θα έχουμε συνεργασία με την μουσουλμανική κοινότητα ή τις κοινότητες που οι περισσότερε από αυτές θεωρούν ότι απειλούνται από τέτοιες ε, πρακτικές γιατί δεν συμφωνούν. Δεν συμφωνούν ούτε συμβάζονται με κάποια παράδοση δική μας εκεί που οι περισσότεροι μουσουλμάνοι προέρχονται από το Μαρόκο όπου τέτοιου είδους συνήθειες δεν συνηθίζονται ούτε είναι τμήμα της παράδοσης. Οπότε θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία με τις μουσουλμανικές αρχές, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την συνεργασία, την συνύπαρξη και την ισότητα των φίλων. Οπότε, για αυτό το λόγο και επαναδιατυπώθηκε το ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους ε, προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων. Αυτό θα γίνει και μέσω της παιδείας. Γι' αυτό σας λέω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό σχετικό το να μπορέσουμε να τονίσουμε το ότι τα περιθώρια δυνατότητες μας δίνει η δική μας ένωμη τάξη μα δίνουν τη δυνατότητα τόσο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, η οποία έχει σχέση με δυσμενεί διακρίσει βάρο των γυναικών, ιδίω στην Ισπανία, λόγω του σχετικού νόμου, του νόμου για την ισότητα. Έχουμε επιφέρει ένα σωρό αλλαγέ, έχουμε κάνει κάποιες τροποποιήσεις ή στον ποινικό κώδικα, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδους επιβολή μέτρων, θέσπιση κάποιων εγκλημάτων, ιδίως σε περίπτωση που παραβιάζεται η ισότητα των φύλων και κατεβλήθη κάποια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική ως προς αυτό, ο, στο, βαθμό που επιτρέπεται από το Ισπανικό δίκαιο και έτσι να μπορούμε να προσθέσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο είδου ειδική ρύθμιση. Διότι μπορούμε να επικαλεστούμε τον ισχύοντα νόμο για να προστατεύσουμε την ασφάλεια, αξιοπρέπεια όλων και ιδίω των γυναικών. Γιατί νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο Σήμερα πρόκειται να περάσει αυτό το μέτρο ή στην ε, Γερουσία και να αυτό κάτι με σύμφωνη. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία υπευλήθησαν σε σχέση με το έργο τη Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω να πω τα εξή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, εν γέννη για όλους μαζί και αν κάτι ξέχασα πρόεδρε ή εσείς να μου το υποδείξετε πρώτα πρώτα και ως παρέθεσαν σου ερωτήματα και πρώτα πρώτα. Τι προβλέπει το πρόγραμμα δράσης για τους ασυνόδευτους ενήλικους. Είναι πρόταση που αφορά αυτό το πρόγραμμα δράσης. Όμως εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης ή στο Λουξεμβούργο πριν από λίγες εβδομάδες. Περιέχει 32 συγκεκριμένα μέτρα. Εδράζοντα σε αυτέ τι αρχέ, σε αυτού του τρει ε, άξονε, του ιδεολογικού σα προανέφερα. Πρόληψη, σχέση με τρίτε χώρε και ανταλλαγή πρακτικών. Διαπίστωση της ηλικίας των λίγων κλπ. Επομένω, ενεκρίθησαν αυτά τα μέτρα και Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε για να δούμε πώς αυτά τα μέτρα θα γίνουν συγκεκριμένες ε, ενέργειες που θα αναλυθούν από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε σχέση με την Frontex. Μάλλον δεν το βλέπουμε τον ε, αποκτήσει καινούργιε αρμοδιότητε Frontex, μάλλον θα πρέπει να γίνει πιο λειτουργική, πιο επιχειρησιακή. Θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να καθίσταται επιχειρησιακή, λειτουργική όσον αφορά τον έλεγχο των ε, συνόρων. Αύριο δε μπορείτε να συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ρούμπα Κλάμπα. Και ένα άλλο ερώτημα που υπευλήθη μπορώ να απαντήσω που αφορούσε την ένταξη. Σήμερα, στη συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει ο κ. Σταβάρες, υπάρχει, λέγω, η νομική βάση ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά την ένταξη. θέματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σαν πολιτικές διακυβερνητικές. Είναι δυνατόν επομένω αυτές οι ενέργειες μπορεί να γίνουν, αυτές οι πολιτικές να γίνουν ευρωπαϊκές. Για θέματα αρμοδιότητας της Ένωσης. Μπορούμε επομένω να έχουμε ως βάση τη στιγμή της Λισαβόνας για να επεξεργαστούμε τέτοιες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ένταξη. Με αυτή την έννοια επομένω, συμφωνούμε με αυτά τα οποία μας είπατε. Όπως τα είπε ο κύριος Θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή την νομική βάση. Μας την παρέχει η συνθήκη. Και σε να κάτσουμε και να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές που μας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε βήματα προόδου σε διάφορους τομείς και όπως είπατε κύριε Μωράες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε εδώ πέρα να καλύψουμε και την ιδέα της ένταξης για το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών αυτό το που σας είπα εγώ συγκεκριμένα ας πούμε όσον αφορά την πολιτική ενόψη του 2020 μια που είμαστε σε μια φάση που έχουμε κάποιες πολιτικές που θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουν δηλαδή την αναδοχή, την υποδοχή των ε, νέων ε, μεταναστών, των νέων αφήξεων, αλλά μιλάμε τώρα για όλο αυτό το τοπίο μιας πλουραλιστικής κοινωνίας που έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, ε, αλλά έχουν την ηθαγένεια κάποιου ευρωπαϊκού κράτους. Επομένως λέμε για τέτοιες πολιτικές οι οποίες ξεκινάνε από την υποδοχή μέχρι να φτάσουμε στη φάση αυτών που ανέφερε ο κ. και, να, και έτσι να μην έχουμε φαινόμενα δυσμενούς διάκρισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω το να προχωρήσουμε έτσι, το να ε, επιτέλεσουμε τέτοιο έργο ε, στο επίπεδο Υπουργών, να γίνει αυτή η ένταξη και ακριβώς αυτό έγινε στη διάσκεψη στην Υπουργή της Αραγώσα για αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα που σας ανέφερα. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε όλα αυτά να τα περάσουμε και μέσα από τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια μέσα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην αποφυγή της μονοδιακρίσεως βάρος μεγάλων μερίδων του ευρωπαϊκού πληθυσμού και να καταλήξουμε σε κάποια συνεκτική κοινωνία που αποτελεί το ευρωπαϊκό μας ε, κοινωνικό πρότυπο. Επίσης, Άκουσε τον προβληματισμό της κυρίας ε, Αντζιβίλ και του κυρίου Μπουσούτρη πάρα πολύ θεμητά αυτά τα οποία διατύπωσαν, μια που έχουμε ασχοληθεί πολύ όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης και προσπαθούμε, να το πω αλλιώς, να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία. Τα δε τελευταία χρόνια νομίζω ότι μπορέσαμε να κάνουμε βήματα πρόοδου, να, να, να συνάψουμε κάποιες συμφωνίες όσον αφορά αυτά τα ζητήματα και έτσι να μπορούμε να έχουμε περισσότερη ομοιογένεια, περισσότερη ε, συνέπεια στις νομοθεσίες τους. Γιατί ακριβώς ήταν θέματα που και εμένα με έκανε πριν από 10 χρόνια. Θυμάμαι η οδηγία για τους προσωρινά εργαζόμενους. Είδαμε ότι έγινε πιο γρήγορη η εκπαιδεύση και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό σε σχέση με την καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση, τη ε, μαύρη εργασία ε, μέσω κάποιων κοινών ε, μηχανισμών για την πολιτική τη μετανάστευση. Επομένω είναι πάρα πολύ λογικό τώρα να μπορέσουμε να δούμε πώ θα ολοκληρώσουμε αυτό το οικοδόμημα, αυτό το κοινοτικό οικοδόμημα να έχει κάποια συνοχή και συνέπεια αλλιώς πώς να κάτσουμε και να, να πολεμήσουμε την ε, παρανομία αν δεν έχουμε περιχαρακώσει αυτή αυτό το, φαινόμενο σε σχέση και με τις αρμοδιότητες της κρατικής των κρατών μελών δηλαδή κάτι το οποίο διατυπώνεται και ορίζεται σαφώς από την θήκη της Λισαβόνας ακόμα βέβαια για το ψηφιδωτό αυτό, λείπουν κάποια κομμάτια. Απασχόληση, προσωρινή απασχόληση. Σας ξαναλέω, δεν άρχισε αυτή η προβληματική, γιατί ακόμα περιμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και με την οδηγία πρόκειται να ρυθμιστεί το θέμα της ε, άδειας και μόνο αυτό που είπε ο κύριο Γιακολίνο θα το καλύψουμε. Πολλέ φορέ ε, ακριβώ είναι πάρα πολύ βάλλοντη θέση αυτών των εργαζόμενων και τον να στη χώρα μα συνδέεται με, κάποια συγκεκριμένη δουλειά, συγκεκριμένη άδεια, συγκεκριμένη δυνατότητα ανέβραση εργασία. Γιατί υπάρχει το Υπουργείο Εργασία και Μετανάστευση. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα θα πρέπει να διαπνέει την ε, οδηγία βέβαια Εξίσου ισχύει το ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο, να υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες για προσωρινή εργασία και άρα να υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ ενός συγκεκριμένου εργαζόμενου και μιας συγκεκριμένης θέσης απασχόλησης. Οπότε, επ' αυτής της βάσης θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση του προβλήματος. Περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν, τόσο ώστε να μπορέσει να μας ε, βοηθήσει και έτσι να συμπληρωθεί αυτό το ψηφιδωτό, αυτό το παζλ. Επομένως, πάρα πολύ ωραία, έχουμε αυτό για την, ε, αυτή την οδηγία και έχουμε και το σχετικό σας ψήφισμα. Μ' αρέσει που το, που το βαφτίσατε ε, με το όνομα του συναδέλφου, του Φέρκας. Ο καθένα θα βάλει το λιθαράκι του για αυτή την υπόθεση. Τώρα, η οδηγία θεωρώ ότι θα πρέπει έτσι να διαμορφωθεί και εμεί προσπαθήσαμε ούτω ώστε να συναυθεί να, συμφωνία και συνένεση στο Συμβούλιο. Να δούμε το πεδίο εφαρμογή, το συζητήσατε. Μπορώ να σας πω ότι προχωρήσαμε προς λιγότερη καταστολή και περιοριστικό πνεύμα όσον αφορά την εφαρμογή, το πεδίο εφαρμογή οδηγία από πλευρά του Συμβουλίου. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσει την ίδια ρότα η Βελγική Προεδρία. Βεβαίω και θα προβούν συνεννοήσει μαζί σας και τελικά ελπίζουμε ότι θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεση τη οδηγία αυτή βεβαίω. και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Και αυτό θα βοηθήσει το να υπάρχει ένα πλαίσιο Συνεπέ για την όλη διαδικασία που ξεκινάει από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, μεταναστών εργαζομένων, που είναι η πλειοψηφία τους άλλωστε. Περιμένουμε από την Κομισιόν να μας κάνει μια πρόταση αξιολόγησης για το τι γίνεται όσον αφορά την μπλε κάρτα. Ελπίζω αυτό θα γίνει σύντομα. Στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας και να δούμε Πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό το μέτρο. Η προσωρινή εργασία, η μπλε κάρτα αφορούσαν και την ε, ερώτηση πώς λέγεστε τρούς. Γιατί είπα για μια συγκεκριμένη περίπτωση, για τους ε, μετανάστες όσον αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα που απασχολεί το Συμβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε είπαμε ότι για την μπλε και για άλλους τομείς της πολιτικής μετανάστευσης εμείς προωθούμε μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαρακτηρίζουν τον αιώνα μας. Και θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο έτσι να διαμορφώνονται οι πολιτικές μετανάστευσης, ε, να δίνουν δυνατότητα κινητικότητας. Και να έχει μετανάστευση το χαρακτήρα εκπαίδευσης, μάθησης, ούτως ώστε αυτό να ισχύει εκεί που πάει κάποιος είτε στη χώρα προέλευση είτε στη χώρα υποδοχής. Και κάποιος να μπορεί να έχει δυνατότητα του να κλείσει τον κύκλο, δηλαδή να γυρίζει από τη χώρα προορισμού στη χώρα προέλευσης. Και η χώρα προέλευσης να γίνεται κάποια στιγμή χώρα προορισμού. Αυτά θα συζητήσει ίσω και αύριο με τον κύριο Ρουμπαλκάμπο όσον αφορά την επανεγκατάσταση. Υπάρχει άλλωστε το πιλωτικό πρόγραμμα της Μάλτας. Θεωρούσαμε ότι είναι τα μέτρα πολύ γενναιόδωρα. Σα αναφέρω δε ότι στην Ισπανία μόλις τώρα θεσπίστηκε νέο νομοθέτημα, ούτω ώστε και εμεί τώρα είμαστε όσον αφορά την επανεκατάσταση. αλληλέγγυη με τις άλλες χώρες γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για υποχρέωση τι τις χώρες και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε αυτούς που έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν, που έχουν περισ... περισσότερους πρόσφυγες, δηλαδή εκεί που υπάρχουν ε, συγκρούσεις, κρίσεις. Βόρεια Αφρική, Ανατολική Αφρική, κάτι τέτοιο είπε την κύριε Κέρκοπ και όσον αφορά τις χώρες από που προέρχονται οι μετανάστες, αυτό είναι πάρα πολύ βασικός άξονας της ε, πολιτικής μετανάστευσης. Είναι τομέας όπου μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδώσει προσθέμενη αξία με τον διάλογο με τις χώρες αυτές. Θα πω στον Αγιοδομήνικο τη Δευτέρα και, και στο Μαρόκο Οπότε, σας λέω αυτό διαρκώς αποτελεί μέλημά μας. Αλλά αυτό αφορά και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα πρέπει να είναι κοινή ευθύνη για αυτό το θέμα, ημών και των τρίτων χωρών. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας, για την παρουσία σας και για την τόσο πλήρη απάντηση στις τόσες ερωτήσεις και ανησυχίες που ακούσαμε. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις ούτε σχόλια, να αποχαιρετήσουμε την κυρία Υφυπουργό για να συνεχίσουμε στην ημερησία διάταξή μας όπως έχουμε προβλέψει. Debería despedirme de estos señores, además. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου ήταν η ευκαιρία που είχα να ξανάρθω. Ε, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Oye,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 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. If you please take your seat. Καθίστε σας παρακαλώ. We get restarted. Ξαναρχίζουμε. As usual, we got a heavy... Ο συνήθως είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη. Ε, ας προχωρήσουμε. Στο σημείο 5 λοιπόν, το οποίο αφορά τον έλεγχο από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε βασικά ψηφοφορία για αυτό το θέμα, που είναι δική μου έκθεση. Ως πρόεδρος της Επιτροπής συνέταξα αυτή την έκθεση μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς τα κράτη-μέλη ελέγχουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αφορά αυτό το άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώην διαδικασία επιτροπολογίας, η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει ξεπεραστεί από τις νέες διατάξεις στο συνθήκη της Αβώνας. Έχω συντάξει έκθεση με τρεις τροπολογίες. Προτείνω ως συζητητής να ψηφίσουμε και τις τρεις τροπολογίες μαζί. Έχει κυκλοφορήσει το σχέδιο της νομοδότησης ε, και καταλόγους ψηφοφορίας. Θα δείτε ότι είναι τρεις ψηφοφορίες. Η μία αφορά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αναφορά που γίνεται σε αυτή. Η δεύτερη αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο ε, Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας. Και η τρίτη ρητά αναφέρει την ανάγκη συμπερίληψης των προπαρασκευαστικών τιμένων. κειμένων. για τις διατάξεις διαφάνειας που αφορούν τα έγγραφα που υπάγονται στον κανονισμό 1049 του 2001. Πριν περάσουμε στη ψηφοφορία, θα πρότεινα να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ο κύριος Μπουσούτηλ ζητεί το λόγο όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα επιθυμούσε να ψηφιστούν χωριστά οι, οι τροπολογίες, συγγνώμη, όχι όλες μαζί. Κυρία Σόμερ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω. Εδώ στα έγγραφά μας έχουμε και ένα έγγραφο του Συμβουλίου. Οι φίλοι της Προεδρίας, τι είναι αυτό, τι ομάδα είναι αυτή, Friends of the Presidency. Θα μπορούσατε να μας επαναλάβετε την ερώτησή σας. Ναι κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτή η, ομάδα Friends of the Presidency Group, οι φίλοι της Προεδρίας. Έχουμε λάβει ένα τέτοιο έγγραφο από το Συμβούλιο. Τι εστί αυτό το πράγμα. Από το Υπουργικό Συμβούλιο. και στο εξώφυλλο γράφει έκθεση της ομάδας φίλων της Προεδρίας. Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι της Προεδρίας, ποια είναι αυτή η ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Σόμερ, μόλις μου λένε ότι είναι μια ομάδα εργασία που συστήθηκε στους κόλπους του Συμβουλίου και φέρει αυτό το όνομα. Friends of the Presidency Group. Εδώ και καιρό εργάζεται. Πρώτη φορά το βλέπω και εγώ μόλις το πήρα είδηση ότι υπάρχει τέτοια ομάδα εργασία που φέρει αυτό το τίτλο. Συμβαίνουν και τέτοια. Καμιά φορά έχει και φίλους η Προεδρία, ξέρετε. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ο κύριος Μισελ, παρακαλώ. Μισελ Μισελ, κύριε Κόπ. Κύριε Κόπ, δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι υπέροχο που η Προεδρία δημιούργησε φίλους. Ίσως πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο πιο φιλικοί απέναντί τους. we should, we should create ναι, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ε, μια ομάδα προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει, ας περάσουμε στην ψηφοφορία τώρα. Όπως πρότεινε ο κύριος Μπουζουτήλ, θα έχουμε χωριστή ψηφοφορία, αφού αυτή είναι η επιθυμία τους. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. said you wanted Νομίζω όλοι έχουμε τις κάρτες μας και θα ψηφίσουμε την κάθε μία τροπολογία χωριστά. Λοιπόν, ψηφίζουμε να κάνουμε πρώτα μια δοκιμή Εντάξει, αυτό είναι μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε ότι όλα λειτουργούν εντάξει. We open a vote. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία τώρα. Όχι. Now we open Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία παριθμών 1. Α, την 3. Ε, Τώρα θα κάνουμε πραγματική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε για τις τρεις τροπολογίες. Τροπολογία 1. Uh, Πρόεδρε, η τροπολογία 1 αφορά αιτιολογική σκέψη και ο κύριος Πουζούτιλ προτείνει να ψηφίσουμε πρώτα τα άρθρα. Επομένως να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες 2 και 3 και η 1 να μείνει για το τέλος. Εντάξει, ξεκινάει η πρώτη ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Now it's 41, 41 plus, 1 minus. 41 υπέρ, μία κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία, όποια και αν είναι αυτή και ό,τι και αναφορά. δεν ξέρω. Εντάξει, την τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία. Και τώρα ψηφίζουμε για την αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 41 υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Final vote. Final vote. Τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Όχι. One missing. Μας λείπει ένας. 21 υπέρ, 2 κατά. 41 υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται. Uh, uh, Περνάμε στο σημείο 6. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικέ υποθέσεις. Έχουμε μια συμφωνία εδώ, η οποία θέτει τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή χρειάζεται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, τον Ονορεύολε Σαλβατόρε Ιακολίνο, να μας παρουσιάσει την έκθεση και εάν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση, ε, καθώς δεν έχει υποβληθεί καμία τροπολογία, θα περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ο κύριος Ιακολίνο έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρόκειται για μια συμφωνία που θα είναι η πρώτη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας Επομένως, υπό αυτή την έννοια, έχει μια ιστορική αξία και μια ιστορική εμβέλεια. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2009, όταν το Ευρωπαϊκό συμφούλιο ε, επέτρεψε τις σχετικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2009 από το ίδιο το Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο ρυθμίζει με πολύ αναλυτικό και ακριβή τρόπο την δικαστική συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγει μια σειρά εχέγγυων εγγυήσεων που πιθανότατα δεν τις βρίσκει κανείς σε άλλες συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν. Υπάρχουν κάποιε προβλέψεις πάρα πολύ σημαντικές που αφορούν τη μετάφραση. Ήδη μας απασχόλησε το θέμα της μετάφρασης. Ε, ήταν ένα θέμα ε, ουσιώδες για την ισότητα, ε, για τις περιπτώσεις ανακρίσεων, προανακρίσεων και και στην ποινική διαδικασία βέβαια. Τώρα εγγυάται η μετάφραση και σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό αυτό. Προβλέπονται επίσης διάφορες διαδικασίες, τηλεδιάσκεψη, καταγραφή εγγράφων, αποσπάσματα και αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών. Μια σειρά ρυθμίσεων λοιπόν που εγγυώνται την αντικειμενικότητα των σχετικών διαδικασιών. Χρήσιμο θεωρώ να αναφέρω ότι ρυθμίζονται όλες οι σχετικές αντιρρήσεις ε, που μπορεί να έχει κανείς στη διάρκεια αυτών των διαδικασιών και που εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία και όλες τις δημόσιες εκφάνσεις, όλες τις δημόσιες πτυχές της συνεργασίας. Υπάρχουν ρυθμίσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και διαδικασίες για άλλα αποδεικτικά μέσα ε, και διάφορες διαδικασίες ε, εγγύησης των δικονομικών ε, θεσμών και διαδικασιών. Ε, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν και πρόσθετα, να συμφωνούν και πρόσθετα μέτρα. Η Ιαπωνία είναι μία από τις ε, παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις μεγάλης σημασίας και η συμφωνία αυτή καταγράφεται ευνοϊκά και από την πλευρά, αντιμετωπίζεται ευνοϊκά και από την πλευρά των Ιαπωνικών αρχών και Χέρι τη στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα μια συμφωνία με τέτοια χαρακτηριστικά που αναγνωρίζει τα σωστά ορθά επίπεδα προστασίας του κατηγορούμενου και του ανακρινόμενου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γραμματεία για τη συνεργασία της, για τη διαθεσιμότητά της. Ε, πρόκειται για ένα έγγραφο που κατά τη γνώμη μου δεν παρουσιάζει Ε, δεν παρουσιάζει σημεία που μπορούν να δεχτούν κριτική. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ευανάγνωστη ε, η συμφωνία. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ιακολίνο. Όπως ανακοίνωσα δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αν δεν θέλει κανένας ευρωβουλευτής και κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρουν το λόγο, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ναι κύριε Μπέιτς. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά εγώ θέλω να προτείνω μια αντίρρηση. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να υπογράφει μόνη της συνθήκες. Και θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ε, το γεγονός ότι το δικαίωμα αυτό είναι εντελώς αθέμητο και παράνομο γιατί δεν παρέχεται ε, δυνατότητα δημοψηφίσματος στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν δύο δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τρία μάλιστα. Η... συνθήκη της Λισαβόνας που είναι 99% ταυτόσιμη με το Σύνταγμα δεν ε, τέθηκε στην λαϊκή ετοιμιγορία και πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι είναι αθέμητο και παράνομο και αντιδημοκρατικό να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να υπογράφει μόνη τη συνθήκε. Και το λέω αυτό γιατί θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Μπάτεν, το είπατε, αλλά αυτό ε, δεν έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου ως Προέδρου να προχωρήσω στην ψηφοφορία γιατί όπως ξέρετε είναι δεσμευτικό δίκαιο η συνθήκη της Λισαβόνας, εφαρμοστέως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας να συνάπτει διεθνείς συνθήκες με άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας και νομίζω ότι πρέπει πανηγυρικά να το δεχτούμε αυτό και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ ορθά δεσμεύτηκε εδώ σε αυτή τη συμφωνία δικαστικής ε, και ποινική συνεργασίας. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα είναι μια ενιαία ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνατε λοιπόν. Ευχαριστούμε για την εργασία σας κυρία Ιακολίνο. Final vote. Τελική ψηφοφορία, εντάξει. Χρειαζόμαστε άλλη μια ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. Τώρα έγινε. We move to point number Περνάμε στο σημείο 7. Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εισηγητής ο κύριος Κοέλιο. Το αντικείμενο, παρακαλώ, Παρακαλώ, συνάδελφοι, σιωπή. Πρέπει να προχωρήσουμε. Το αντικείμενο είναι η εξέταση της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης και η παρουσίαση της γνωμοδότησης της Νομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Επίσης, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Στα επόμενα λεπτά λοιπόν ο κύριος Κοέλιο θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης για την τροποποιημένη πρόταση για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ασχοληθούν με το ζήτημα το οποίο τέθηκε σε αυτού. Σας θυμίζω, το Ευρω... η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας ρώτησε εάν η ίδρυση αυτού του οργανισμού που θα είναι υπεύθυνο για το SIS-2, για το VIS και το Eurodac, πρέπει να βασιστεί σε ένα ή σε περισσότερα νομικά έγγραφα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν σε όλα αυτά τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα ή δεν συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές ενός πληροφοριακού συστήματος και η Ισπανική Προεδρία ε, μπορεί να σχολιάσει πάνω σε αυτό, μπορεί να κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό ε, και θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να παρέμβουν και αυτοί. και εμείς παρεμβαίνουμε και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα σοβαρό νομικό πρόβλημα για αυτήν την έκθεση. Και μέχρι στιγμής ε, η συνάντηση της Προεδρίας με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και οι δύο κύριες χώρες, το Βρετανικό, η Βρετανία και η Ιρλανδία, θα ξεκινήσουν, ε, θα έρθουν εδώ στις 11 και 4. Το ξεκινάνε τώρα, τελειώνει τώρα η συνάντησή τους. Πρέπει να τους περιμένουμε γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μας και τα σχόλιά μας και αυτά θα μείνουν αναπάντητα. Πρόεδρος. Εντάξει, θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό και θα αναβάλουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης μέχρι να λήξει η συνάντηση που αναφέρατε. Επομένως, προτείνω να αναβάλουμε για ένα τέταρτο, να διακόψουμε για ένα τέταρτο τη συνεδρίασή μας. Λοιπόν, να είστε πίσω σε ένα τέταρτο. Ευχαριστώ. δεν

Uh, Κύριοι συνάδε... αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ήρθε ώρα να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Παρακαλώ καθίστε. We have... Uh, ε, σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης ε, ίδρυση και λειτουργία ενός οργανισμού για μεγάλα συστήματα πληροφορικής στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, πρώτα ο συνάδελφος Κάρλος Κόέλο θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης, μετά θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της νομικής υπηρεσίας για το θέμα που προέκυψε για το κατά πόσο η ίδρυση αυτού του οργανισμού που θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργική διαχείριση του SIS-2, και Eurodac θα βασίζεται σε ένα ή σε περισσότερα νομικά έγγραφα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα σχόλια της Προεδρίας για το συγκεκριμένο ζήτημα και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν θέλουν να παρέμβουν και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση για, την, για το σχέδιο έκθεσης. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα σχετικά με αυτόν τον οργανισμό. Ένα νομικό πρόβλημα και ένα πρόβλημα ουσίας. Και νομίζω ότι πρέπει να χωρίσουμε τη συζήτηση. Διαφορετικά θα είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που σας προτείνω λοιπόν είναι να δώσουμε το λόγο τώρα στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, να ακούσουμε την απάντηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής αν θέλει να δώσει μια απάντηση. Γιατί, Γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το αν θα έχει μια ενιαία πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλούμε για έναν οργανισμό που θα διαχειρίζεται διαφορετικά συστήματα όπου τα δικαιώματα συμμετοχής των ε, κρατών μελών διαφέρουν. Για παράδειγμα, η Βρετανία δεν συμμετέχει στο ΒΙΣ ούτε στο ΣΥΣ παρά μόνο σε ένα μικρό κομμάτι του. Και ενώ συμμετέχουν πλήρω, συμμετέχει πλήρω η Βετανία στο σύστημα Eurodac. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα μεταβλητή γεωμετρία και ένα τεράστιο νομικό πρόβλημα όσο αφορά την υιοθέτηση αυτή της πρωτοβουλία. Προτείνω λοιπόν πρώτα να ασχοληθούμε με το νομικό ζήτημα να ακούσουμε την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και την απάντηση του Συμβουλίου και την απάντηση της, Επιστροπή, Επιτροπής και στη συνέχεια να παρουσιάσω την ουσία της έκθεσής μου και να ακολουθήσει η συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κουέλο. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στους εκπροσώπους της νομικής υπηρεσίας να προσπαθήσουν να απαντήσουν το ερώτημα. Thank you. Ευχαριστώ ευχαριστούμε για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την γνώμη της Νομικής Επιτροπής επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οργανισμό αυτό που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση τριών συστημάτων του ΣΥΣ, δύο του ΒΙΣ και του ΓΙΡΟΝΤΑΚ. Και όπως είπε ο εισηγητής, το νομικό πλαίσιο αυτών των ε, συστημάτων περιπλέκεται από το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα ή σε όλες τις συνιστώσεις τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συμμετέχουν πλήρως στο Eurodac, το οποίο δεν έχει να κάνει με τα κεκτημένα του Σέγγεν, δεν συμμετέχει καθόλου στο ΒΙΣ, συμμετέχει εν μέρη στο ΣΥΣ2 με βάση τη συμμετοχή στα κεκτημένα του Σέγγεν. Το θέμα είναι κατά πόσο η ίδρυση του οργανισμού πρέπει να βασίζεται σε ένα ή σε περισσότερα νομικά έγγραφα. Υπήρξε μια υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την άρνηση του Συμβουλίου να επιτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στην έγκριση του κανονισμού ε, ε, για το Frontex. Το Συμβούλιο αρνήθηκε επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε σε εκείνο το μέρος του κεκτημένου που αφορούσε τους νοριακούς ελέγχους. Το, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο προσέφυγε με αγωγή κατά της άρνησης του ε, Συμβουλίου και το δικαστήριο είπε ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εξελίξεις του κεκτημένου αν δεν συμμετέχουν σε αυτό για παράδειγμα στην πολιτική θεωρήσεων ή στους συνοριακούς ελέγχους. Στην πρόταση του η Επιτροπή συμπεριέλαβε μια σειρά αιτιολογικών σκέψεων που αντικατοπτρίζουν τους περιορισμούς της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Αυτό συνάδει με την νομολογία. Στο 24 σημείο λέγεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έγκριση και στη συνέχεια λέει το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στην έγκριση. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει για την Ιρλανδία. Αυτές οι αιτιολογικές σκέψεις ε, είναι αντιφατικές. Δηλαδή, είτε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συμμετέχουν στην υιοθέτηση όλου του κανονισμού ή όχι. Αν τους επιτροπεί να συμμετέχουν στην έγκριση του κανονισμού, τότε θα πρέπει να συμμετέχουν σε μέρη που είναι μεταξέλιξη του κεκτομένου που δεν έχουν αποδεχθεί, στο οποίο δεν συμμετέχουν. Πρέπει να ε, υπάρξει συνοχή με, το, με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. αλλιώς θα προκύψει νομική αβεβαιότητα. Θα πρέπει να διασαφινιστεί το ποσοστό συμμετοχής της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ζήτημα όμως, εάν μπορούν να συμμετέχουν στη ψηφοφορία του κειμένου συνολικά, παραμένει ανεπίλητο. Ε, θα υπάρξει Υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής των χωρών αυτών σε συγκεκριμένα τμήματα του εγγράφου, αλλά αυτό προκαλεί πολιτικά προβλήματα. Προτείνεται και μια άλλη λύση, αλλά θα αφήσω το Συμβούλιο να την εξηγήσει. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την άποψη της Ισπανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα καταλάβατε από τα όσα είπε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, το θέμα δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι λίγες ε, οι συνεδριάσεις, ούτε η ανησυχία που προκάλεσε στο Συμβούλιο αυτό το θέμα. Καθυστερήσαμε λίγο να φτάσουμε στη συνεδρίασή σας, γιατί εργαζόμαστε ακριβώς επ' αυτού με τα ε, κράτη-μέλη ε, που θίγονται και την Προεδρία. Δεν θα σας κουράσω γιατί θεωρώ, δεν θεωρώ ότι έχω εξουσιοδότηση να μιλήσω νομικά. Θα αφήσω την εξήγηση της πιθανής λύσης που μάλλον ε, βρέθηκε από πλευρά Συμβουλίου να ε, εκφραστεί ε, από μια εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας που παρευρίσκεται. Thank Um, Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να προτείνουμε μια λύση. Τη λύση την οποία σκεφτήκαμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Πράγματι, συμφωνούμε με την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν ε, επιπλοκές ε, σε σχέση με την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στην πρόταση για τον Οργανισμό Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων για τους λόγους που εξηγεί η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρεί, εξετάσαμε επίσης την δυνατότητα ε, να διαιρέσουμε την πρόταση στα δύο, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαιρεθεί η πρόταση σε πολλά μέρη. Για πολλούς και διάφορους λόγους και για πρακτικούς λόγους, καθώς το όπως εξήγησε η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν τέλει είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Αφού σκεφτήκαμε όμως ως προς το πώς θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς να διαιρέσουμε την πρόταση, καταλήξαμε σε μια άλλη λύση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλου στα κεκτημένο του Σέγγεν. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλου του κεκτημένου του Σέγγεν, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν ανα πάσα στιγμή να ζητήσουν να συμμετέχουν σε όλο ή σε μερικές διατάξεις του κεκτημένου του Σέγγεν. Τώρα, σχετικά με την πρόταση για τον Οργανισμό Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, θεωρούμε ότι αυτό είναι δυνατόν, γιατί πράγματι είναι μια πολύ ειδική περίπτωση γιατί αφορά όλα εκείνα τα μέρη όπου το Ηνωμένο Βασίλειο και η ή δεν συμμετέχουν ή συμμετέχουν εν μέρη, ε, η λύση θα μπορούσε να είναι να ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και η να συμμετάσχουν στην υιοθέτηση της πρότασης επί τη βάση του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου του Σέγγεν και το Συμβούλιο θα αποφασίσει ομόφωνα θα εξετάσει το αίτημα αυτό της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα αποφασίσει ομόφωνα. Θα είναι απόφαση του Συμβουλίου παρόμοια με την ε, απόφαση 2365 όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε να συμμετέχει σε ορισμένες πτυχές του κεκτημένου του Σέγγεν και τότε το Συμβούλιο το επέτρεψε αυτό, επέτρεψε στην Ιρλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχουν εν μέρη στο κεκτημένο του Σέγγεν. Αυτή θα μπορούσε να είναι η λύση. Και με αυτή τη λύση το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να συμμετέχουν πλέον στην έγκριση των προτάσεων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων συνολικά. Ήδη ενημερώσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για τη λύση αυτή. Και μέχρι στιγμής ε, η απάντηση από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θετική και λένε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα, θα υποβάλει αυτό το αίτημα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Θα ζητήσει λοιπόν να συμμετάσχει στην ε, έγκριση του κανονισμού συνολικά Προς το παρόν η Ιρλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτημα. Αφού λάβουμε αίτημα από μία ή από τις δύο αυτές χώρες, τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιτρέψει στις χώρες αυτές να συμμετέχουν στην έγκριση του κανονισμού συνολικά. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι η... μια έγκυρη νομική λύση για το πρόβλημα και δεν θα υπάρχει πια ανάγκη να διαιρεθεί η πρόταση σε πολλά μέρη. Ενώ την, πρόταση για την εγκαθίδρυση και την λειτουργία του οργανισμού θα παραμείνει ως έχει. Οι αιτιολογικές σκέψεις θα παραμείνουν ως έχουν και θα αποφύγουμε τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να λάβουν το λόγο. Θέλουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια από αυτές τις περιπτώσεις που όλοι συμφωνούν με τα γεγονότα και τις παραδοχές, αλλά πρέπει να βρούμε τις λύσεις για να ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές και τα γεγονότα. Ακούσαμε τις προτάσεις ε, των νομικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, είναι θέμα μεταβλητής γεωμετρίας, είναι υβριδικό ζήτημα όπως λέγεται. Ωστόσο το υπάρχει, το προηγούμενο, ε, ήδη έχουμε αντιμετωπίσει μια νομική πράξη με τέτοια μεταβλητή γεωμετρία και γι' αυτό η Επιτροπή πιστεύει με βάση όλα τα στοιχεία ε, ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ενιαίο το κείμενο με τις απαραίτητες διασαφηνίσεις για το πεδίο εφαρμογής και τους διάφορους τύπους συμμετοχής των κρατών μελών ως προς τα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την υβριδική κατασκευή. Ε, μια, ένα και ενιαίο κείμενο είναι η σωστή λύση. Γιατί, Γιατί αν μοιράσουμε τα έγγραφα θα μην διαιρώντας τα κείμενα επιτυγχάνουμε ένα καλύτερο πνεύμα ρυθμιστικό και υπηρετούμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας επί τη βάση όλων των τροπολογιών και των αναπροσαρμογών και των προσταφερέσεων που έχουμε κάνει στα νομικά κείμενα. Επίσης πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Αν διαιρέσουμε τα κείμενα και πάλι θα καταλήξουμε σε υβριδική κατασκευή όσο αφορά αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Γιατί το πιο περίπλοκο κομμάτι της μεταβλητής γεωμετρίας δεν αποφεύγεται. Ακόμα και αν χωρίσουμε το Eurodac από το VIS, που είναι σαφής η συμμετοχή των μερών, όσο αφορά το SIS 2, πάλι θα έχουμε αυτή τη μεταβλητή γεωμετρία. Γι' αυτό λοιπόν, διαρώντας τα κείμενα, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Πάλι καταλήγουμε σε μια υβρίδικη κατασκευή, τουλάχιστον για αυτές τις δύο χώρες και το σύστημα ΣΥΣ-2. Και θα έχουμε πάλι πολλές νομικές πράξεις αντί για μία, πράγμα που περιπλέκει το νομικό πλαίσιο. η γλώσσα που επιλέξαμε αν θα προσέξετε την ανάγνωση των αιτιολογικών σκέψεων 24 και 25, θα δείτε ότι λέγεται εκεί, γιατί με μεγάλη προσοχή συντάξαμε αυτές τις παραγράφους, λέει εκεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα συμμετέχουν στην, στην έγκριση του κανονισμού παρά μόνο στο μέτρο που. Έχουμε αυτό την έκφραση στο μέτρο που που πιστεύουμε καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, την έκταση εφαρμογής του νομοθετήματος στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, και σίγουρα θα ήμασταν ευτυχείς μαζί σας να βρούμε και μια πιο σαφή διατύπωση, να, δια... Υπάρχει επίσης και ένα άλλο ζήτημα. Ένα ζήτημα δικαιοσύνης θα έλεγα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συμβάλλουν οικονομικά στην ε, λειτουργία του οργανισμού όπως όλες οι άλλες χώρες. Το γεγονός λοιπόν ότι συμμετέχουν σε ορισμένα από τα συστήματα που θα διαχειρίζεται αυτός ο οργανισμός πιστεύω ότι τους, δίνουν τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής και της ψηφοφορίας παρόλο που, όπως λέγεται, σαφώς στο προήμιο αυτό δεν θα βλάψει την συμμετοχή στις ψηφοφορίες και τη γενική λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, καταγράψαμε και τη λύση που προτείνει τώρα το Συμβούλιο, η νομική του υπηρεσία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βρούμε μια επικοδομητική ε, λύση για να αποφύγουμε αυτή την περίπλοκη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι ότι είναι κάτι πολύ καινούργια αυτή η πρόταση και αναμένουμε την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Θα, θα δω λοιπόν πώς θα αποκρισταλωθούν οι απόψεις των χωρών αυτών και στη συνέχεια θα προσπαθούμε να βρεθούμε μαζί με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για να βρούμε τη σωστή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάρλος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική μας υπηρεσία για τη σαφήνεια της νομοδότησής της και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βρήκαν από τη φαίνεται λύση και στο Συμβούλιο για να επιλύσουν το νομικό πρόβλημα και ελπίζω και η Ιρλανδία να ενταχθεί όπως ζήτησε και το Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δημιουργήσουμε τον οργανισμό αυτό. Θα ήθελα να σας προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, 12 Ιουλίου, ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, εξ όσο γνωρίζω η έκθεσή μου υπάρχει ήδη σε όλες τις γλώσσες. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω 8 σύντομα σημεία. Πρώτον, γιατί χρειαζόμαστε οργανισμό διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει με τρόπο επίσημο και τυπικό μια τέτοια μορφή οργανισμού. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους η αρμοδιότητα δεν θα πρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε η ίδια Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν έχει τα μέσα ούτε τη θέληση να κάνει κάτι τέτοιο. Και ο εκτελεστικό οργανισμός επίσης δεν είναι λύση. Για ποιο λόγο. Διότι το κοινοβούλιο, το, το δεν μπορεί να ελέγχει δημοκρατικά με τον ίδιο τρόπο ένα τέτοιο οργανισμό και δεν μπορεί να διαμορφώνει ε, τον οργανισμό ε, παρά μόνο αν είναι ευρωπαϊκός. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός λοιπόν, η agency είναι η καλύτερη λύση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα νέα συστήματα, νομίζω ότι Εάν ο οργανισμός αυτός είναι αρμόδιος για νέα συστήματα προφορικής, αυτό θα πρέπει να έχει κάλυψη νομική, δηλαδή με νομικά μέσα, με συναπόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί με τρόπο σαφή στο κείμενο. Τρίτον, νομίζω θα πρέπει να διευκρινίσουμε τους στόχους και τα καθήκοντα του οργανισμού αυτού. Άλλωστε έχω κάνει και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Σημείο τέταρτο. Τα διάφορα έργα που θα αναλαμβάνει θα πρέπει και πάλι να έχουμε θεσπίσει κανόνες για να μην ε, έχουμε πιλωτικά προγράμματα που de facto να πολλαπλασιάζουν και να διευρύνουν το πεδίο που καλύπτει ο οργανισμό αρμοδιοτήτων. Έχω κάνει λοιπόν προτάσεις και πάλι με τροπολογίε για να καλύπτονται τα ε, πιλωτικά προγράμματα. Η έδρα τώρα είναι το πέμπτο θέμα. Έχουμε προτάσεις ε, δύο από τη ε, Εστονία συγγνώμη, και από τη Γαλλία. Το Κοινοβούλιο από νομικής πλευράς δικαιούται να αποφασίζει σε ίσους όρους με το Συμβούλιο. Γιατί είναι στην απόφαση είπαμε. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια παράδοση ε, για την έδρα να το αποφασίζει το Συμβούλιο. Εμεί δεν θα διαπλεκτιστούμε γι' αυτό. Εάν το Συμβούλιο προτείνει μια καλή λύση, δεν θα είναι το Κοινοβούλιο εκείνο που θα την εμποδίσει ή θα την αντικρούσει. Θα πρέπει όμως να δώσουμε και κάποιες παραμέτρους, ε, όρους και προϋποθέσεις, αν θέλετε, για να βοηθήσουμε το Συμβούλιο να λάβει την απόφαση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μερικές ε, τροπολογίες και πιστεύω πώς να το πω, ε, να βελτιώσουμε κάπως τα πράγματα. Σημείο έκτο και τελειώνω σιγά σιγά. Υποδομή της επικοινωνίας. Εγώ δεν είμαι κατά της ιδέας να ε, έχουμε εξωτερικές αναθέσεις για την υποδομή αυτή, αλλά και πάλι με όρους και προϋποθέσεις. Για ε, να τα δίνουμε με τρόπο σωστό, με διαγωνισμούς. Και πάλι έχω κάνει τέτοιες τροπολογίες. Έβδομον. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιώματα ψήφου. Όπως θα έχουμε όλοι καταλάβει σήμερα, ε, είναι διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα τα δικαιώματα ψήφου. Αν μια χώρα δεν δεσμεύεται από, πώς να το πω τώρα, ε, νομικά συστήματα θα πρέπει να έχει δικαίωμα να λαμβάνει διαβαθμισμένες πληροφορίες, να συμμετέχει στη συζήτηση και στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή, το δικαίωμα συμμετοχής και το δικαίωμα ψήφου ε, θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με τη συμμετοχή των διαφόρων κρατών μελών στα συστήματα. Ο πρόεδρος, κατά τα άλλα πιστεύουμε, του οργανισμού αυτού θα πρέπει να επιλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη και εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη εκείνα που εφαρμόζουν πλήρως ε, ε, όλους τους κανονισμούς και είναι πλήρη μέλη εκεί. Δεν έχει νόημα δηλαδή ο πρόεδρος να είναι ε, από ένα κράτος μέλος που δεν συμμετέχει πλήρως παρά μόνο μερικά στη διαδικασία αυτή. Τελευταίο, 8. Προστασία δεδομένων και δημοκρατικός έλεγχος. Έχω κάνει και εκεί πολλές τροπολογίες έτσι ώστε να έχουμε υψηλότερη προστασία δεδομένων, δημοκρατικό έλεγχο και με τη βοήθεια των συναδέλφων ελπίζω να έχουμε καλύτερε απολογίε μέχρι τι 12 Ιουλίου, σα είπα στι 12 το μεσημέρι, για να μπορέσει να συζητήσει στη συνέχεια και να ψηφίσει μετά τι ελληνές διακοπέ το Σεπτέμβριο η Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατα, λέει η Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Κουέγιο. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση. Uh, Έχουν ζητήσει το λόγο δύο μέλη τη επιτροπή μα, ο κύριος Άρμπρεχτ και η κυρία Λάτσφορτ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Καλώς. Ορίστε κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Κάρλος Κουέλιο για την έκθεσή σου. Χαιρετίζουμε αυτές τις τόσο εύστοχες τροπολογίες. Και επίσης αυτές τις επικρίσεις όσον αφορά την, και τον κατευθυνόμενο υποδομή για τις βάσεις δεδομένων και για την προθέση των δεδομένων θέλω να σας πω ότι αυτές οι διατάξεις κατά της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων είναι σε μια κλειδί για το Κοινοβούλιο. Επίσης εξεκαθαρίζουμε ότι αυτό θα είναι μεγάλη σημασία για μας και για το μέλλον. Οπότε όχι, δεν έχουμε τώρα μια εναλλακτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, αυτήν όλη την υποδομή και να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στην διαλειτουργικότητα. Όμως, είναι θεμέλιος λήθος για την υπόθεση αυτή κατά τη γνώμη σου δεν θέλουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο λόγω της προστασίας των δεδομένων γιατί διαπιστώνουμε κάποιους κινδύνους που ενεδρεύουν όσον αφορά κάποιες βάσεις που έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους. Επομένως, γι' αυτό και δεν θέλουμε να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Έτσι βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Αλλά να μην έχουμε κάποιες θετικές κατηγορηματικές διατάξεις σχετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα και ίσως και για το κοινοβούλιο γενικότερα να κάνουμε μια τέτοια ρύθμιση. Γιατί αυτό θα απασχολήσει έντονα την Επιτροπή μας. Κυρία Λάντφορντ, Βαρόνι ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Άλμπλεχτ. Ανέκαθεν με μεγάλη προσοχή στην Επιτροπή μας ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και επίσης προσωπήθηκε από τον κύριο Κοέλιο για το ότι το να υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, με τέτοια συγγνώμη οργάνωση δεν σημαίνει ότι έχουμε τις εγγύησεις που προσφέρει η διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι διαφορετικό θέμα και θεωρητικά ακόμα. Πρόκειται για διαφορετικά πράγματα επομένως. Γιατί να μην υπάρχουν τέτοιες έμεσες συνέπειες από την ε, διαχείριση την κοινή, εάν γκρεμίσουμε τους τείχους, το συνικό τείχος λέω που χωρίζει τις διάφορες βάσεις δεδομένων. Πάρα πολύ αξιόλογη η δουλειά του κ. Κοέλιο, άλλωστε έχει μακρά εμπειρία για το SIS και για τη διαχείριση των βάσεων αυτών δεδομένων. Άρα χρειάζονται κάποιες εύστοχε διατάξεις, ώστε να έχουμε καλή προστασία, καλή διαχείριση και τήρηση των κειμένων διατάξεων για αυτή την περίπτωση τώρα. Για Αμερικανής δεν έχω διαβάσει ούτε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και επειδή άργησα να έρθω δεν άκουσα και τι είπε και προβλέπει τι ανέπτυξε η υπηρεσία του Συμβουλίου. Πάντως, ο Κάρλος Κοέλιο νομίζω ότι προτίθεται να λάβει υπόψη ότι σοφό προκύψει από τις ε, επαφές με το Συμβούλιο, βέβαια εντός κάποιων ορίων, γιατί έχει δίκιο ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε οι μη συμμετέχουσες χώρες να υπερβούν τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στα δικαιώματά τους όσον αφορά την προσβασιμότητα στο SIS. την πρώτη μορφή του SIS τέλο πάντων. Το ίδιο σχέδιο για αυτούς που δεν συμμετέχουν στην Eurodac. Το ότι η κυβέρνηση έγινε αντιπολίτευση δεν αλλάζει την απόψή μα όσον αφορά την ε, δέουσα τήρηση αυτών των ορίων που τάσει ο νόμος. Έχουμε άλλωστε και την ομολογία του δικαστηρίου όσον αφορά τη Frontex, αυτές τις βάσεις δεδομένων, νομολογία που οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Εξαρτήτως τάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, φυσικά και νομιμοποιούνται όλοι να προσπαθούν να πετύχουν όσο γίνεται καλύτερες λύσεις. Ελπίζουμε ότι η σαφήνεια θα επιτευχθεί και θα υπάρχει μια σφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση με διαφοροποιημένες ρυθμίσεις που θα υπάρχουν και θα διέπονται από διαφάνεια και έτσι δεν θα επιφέρουν κάποια σύγχυση για το μέσο χρήστη. Τώρα με τη Συνθήκη Λισαβόνα ελπίζουμε ότι ένα πλεονεκτήμα δεν είναι, θα υπάρχει κάποια ενωπημένη αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων. Πάντω η τελική ρύθμιση του από τι θα διέπεται, ποιο θα δικαιούται να έχει πρόσβαση, αυτό πρέπει να είναι μια ρύθμιση σαφής, ξεκάθαρη. Ακρίβεια σφαιρική αντιμετώπιση που ελπίζουμε ότι μεταξύ τους είναι συμβατά και έτσι μπορούμε κάπου να καταφέρουμε όσον αφορά τα όρια που δεν μπορεί κανείς να υπερβεί εάν δεν συμμετέχει. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες ας πούμε ασφαλιστικές δικλείδες που μας παρέχει το, το, το κεκτημένο του Σέγγεν. Ποιο ξέρει, ίσως ε, για μερικά χρόνια ακόμα πρέπει να περιμένω τόσο ώστε να γίνει η ελπίδα για πραγματικότητα για την Ιρλανδία, τη χώρα μου κλπ. Σα. ευχαριστούμε κύριε πρόεδρο. Τώρα, μπα και θέλει η Προεδρία να λάβει το λόγο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι για την Ισπανική Προεδρία ασχοληθήκαμε το τελευταίο εξάμεινο με επιτυχία ή λιγότερη επιτυχία με το θέμα αυτό μετά από τη Σουηδική Προεδρία και με χαρά βλέπουμε ότι αρχίζουν να αποκρισταλώνονται κάποιες απόψεις στο κείμενο που έχει συζητηθεί σε ομάδες εργασίες και είναι πολύ μεγάλη η ευθυγράμμιση πλέον με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειαζόταν να επιμείνω εγώ σε κανένα από τα σημεία γιατί με θαυμάσιο τρόπο το εξέθεσε ο κύριος Κοέγια. Εργάζεται το Συμβούλιο στα σημεία αυτά και ήδη η πλειοψηφία είτε έχει συμφωνήσει είτε έχει αναγνωρίσει ότι είναι περίπλοκα και θα τα μεταφέρει σε πολιτικό επίπεδο για λήψη απόφασης. Υπό την έννοια αυτή Κυρία Πρόεδρε, το παραπέμπουμε πλέον στο επίπεδο των πολιτικών του Συμβουλίου. Θα ήθελα να πω το εξή τώρα στα δύο μέλη του Κοινοβουλίου που μίλησαν εκτό από τον κύριο Κολέγιο. Θα ήθελα να σα διαβεβαίωσω και να σα δώσω τα μέγιστα εχέγγυα και από πλευρά τη Ισπανική Προεδρία αλλά και Συμβουλίου γενικότερα ότι στη δημιουργία του οργανισμού αυτού κανένα δεν θέλει να παραβιάσει τα νομικά συστήματα, τις νομικές βάσεις, ούτε κατά διάνοια. Το κάθε τεχνικό κείμενο ορίζει τις λεπτομέρειες τις νομικές και όταν θα σε ισχύ και τα, νομικά ε, ε, τα πιλωτικά προγράμματα και τα συστήματα, τα μελλοντικά θα λειτουργούν σωστά. Πάντως, Χρειάζεται για να λειτουργήσει ο οργανισμός αυτός ε, μια νομική βάση, ένα νομικό κείμενο, συμφωνία κοινοβουλίου του Συμβουλίου. Είναι γνωστά αυτά τα θέματα, είναι συνηθισμένα και με κάθε μετριοφροσύνη σας εγγυώμαι από πλευρά της Ισπανικής Προεδρίας ότι όλα θα λειτουργήσουν σωστά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα η Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή για την έκθεση και το πολύ επικοδομητικό έργο που έγινε. Πράγματι, αν δείτε όλες τις τροπολογίες, η τεράστια πλειοψηφία τους είναι αποδεκτή. Στην Επιτροπή είτε ως έχουν, είτε με ίσονο σημασίες αναδιατυπώσεις. Ένα μικρό παράδειγμα. Καλωσορίζω όλους ιδιαιτέρως ε, τις υποδείξεις ε, για τη διαδικασία διορισμού ε, του διευθυντή. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες τροπολογίες και παραδείγματα όπου πιστεύουμε πως η προτάσεις της έκθεσης πραγματικά ενισχύουν το κείμενο όσο έχει. Αυτή είναι, αυτό είναι το γενικό σχόλιο, ο γενικός τόνος της θέσης μας. Επιτρέψτε μου τώρα να θίξω κάποια ζητήματα πάνω στα οποία έχουμε ανησυχίες για τη διατύπωση. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ γρήγορα να τα καλύψω. Καταρχήν, το ζήτημα της υποδομής επικοινωνιών. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα στο ζήτημα αυτό. Ε, οι διαχειριστικές όψεις του συστήματος σίγουρα υπάρχουν στην νομική βάση όλων των συστημάτων ε, και υπάρχει ειδική μνήα στο κείμενο. Ε, αυτή η μνήα δεν μπορεί παρά να διευκρινίζει και να ενισχύει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Ωστόσο, αναφέρομαι στην τροπολογία 14. Πιστεύουμε ότι οι αναλυτικές συνθήκες και όροι που περιέχονται σε αυτή την τροπολογία υπερβαίνουν το μέτρο του απαραίτητου. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί ήδη στη νομική βάση κάθε συστήματος, του ΣΥΣ2, του ΒΙΣ και του ΓΙΡΟΝΤΑΚ, έχουμε σαφείς όρους και προϋποθέσεις για την ασφάλεια των υποδομών επικοινωνίας των δικτύων, και οι όροι και συνθήκες υπάρχουν ήδη εκεί. Δεν, δεν έχει νόημα να περιπλέκουμε ή να συμπληρώνουμε ε, αυτές τις προϋποθέσεις. Επιπλέον οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τόσο των ε, συμβατικών όψεων όσο και των ε, όψεων ασφάλειας θα παραμένουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του οργανισμού, για το ΣΥΣ2 για παράδειγμα. Και γι' αυτό, σε αυτό το κείμενο για την ίδρυση του οργανισμού να περιληφθούν προϋποθέσεις και όροι για τις επικοινωνίες, για την για τις υποδομές, τις επικοινωνιακές και την ασφάλεια δεν έχει νόημα γιατί αυτό θα παραμείνει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, όπως είπα και πριν. Επίσης, ε, η λεπτομερής περιγραφή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων νομίζουμε ότι ε, προσωμιάζει με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ενός ε, διαγωνισμού. Όπως είπα και πάλι αυτό θα παραμείνει στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δεν έχει νόημα να περιγράφονται με, τέτοια, με τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας. Ένα άλλο σχόλιο, η τροπολογία 24 που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει λόγος που προτείναμε δύο μέλη αντί για ένα και γιατί στο συγκεκριμένο οργανισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν ρόλο που υπερβαίνει τη συνήθι θεσμική της συμμετοχή σε τέτοια διοικητικά συμβούλια. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατηρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την υποδομή των επικοινωνιών, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πάνω από, το, πάνω από μια θέση που συνήθως έχουμε. Και γι' αυτό το προτείναμε αυτό και θέλουμε να επιμείνουμε στην πρότασή μας να έχουμε δύο εκπροσώπους στο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Όσο αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για τα για ε, τροπολογίες 13 και 14 για τις χώρες που δεν συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές των πληροφοριακών συστημάτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η μεταβλητή γεωμετρία συμμετοχής. Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι κάτι που δεν πρέπει να ακολουθεί αναγκαστικά την ίδια λογική γιατί όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον οργανισμό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, σε αυτές τις πληροφορίες, ακόμη και αν δεν έχουν δικαίωμα ψήφου πάνω σε αυτά. Πιστεύουμε ότι τα περισσότερα ζητήματα θα απλώνονται εγκάρσια στις δραστηριότητες του οργανισμού. Θα έχουν σχέση ε, με τη διαχειριστική πλευρά που θα αφορά όλα τα ζητήματα. Επομένω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε κατά πόσο ένα κράτος μέλος θα μπορεί να βλέπει μέρη μόνο ενός εγγράφου, ενώ δεν θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο έγγραφο. Νομίζουμε ότι αυτό θα περιέπλεκε τα πράγματα και δεν υπάρχει και λόγος. Για τις συμβουλευτικές ομάδες. Εν ολίγης πιστεύουμε ότι η λογική του να έχει κανείς συμβουλευτικές ομάδες είναι να έχει το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ε, λόγω και της έκτασης και του εύρους των συστημάτων αυτών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια προσθήκης και άλλων συμβουλευτικών ομάδων σε περίπτωση που επεκταθεί η αρμοδιότητα του οργανισμού και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ως προς τη δημοσίευση τώρα της διαδικασίας επιλογής για τον εκτελεστικό διευθυντή, σύμφωνα με τις τροπολογίες του εισηγητή, που προτείνεται αυτό να γίνει μετά από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς προτείνουμε να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός, γιατί είναι προς το συμφέρον της ταχείας ε, σύστασης του οργανισμού να, να μπορεί να δημοσιεύσει να διαφημίσει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή ακόμα και πριν από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς, καθότι έχουμε την ευθύνη της προκήρυξης αυτών των θέσεων, θα ήμασταν πρόθυμοι να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες τις σχετικές πριν από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, ε, για τα δικαιώματα ψήφου των συνδεδεμένων μελών, σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαμε με το Συμβούλιο, προσανατολιζόμαστε στο να αφήσουμε τα ζητήματα δικαιώματος ψήφου ε, για την περίοδο διαπραγμάτευσης της συμμετοχής των συνδεδεμένων μελών στον οργανισμό. Δεν θα θέλαμε να, συμμετέχουμε, να, συμπεριλάβουμε τα δικαιώματα ψήφου στο κείμενο, γιατί αν τα, γιατί αν τα συμπεριλαμβάναμε στο κείμενο, τότε θα θεωρεί το ελλείψη άλλης ρύθμιση ότι Ήδη έχουν δικαιώματα ψήφου οι χώρε αυτέ, ενώ αυτά τα δικαιώματα ψήφου πρέπει να συζητηθούν κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων των συμφωνιών σύνδεση. Τέλο, για την διαλειτουργικότητα θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι κάτι που πάντα απασχολεί την Επιτροπή, το βλέπει με μεγάλη προσοχή. Υπάρχει η νομική βάση κάθε ενός από αυτά τα συστήματα που ορίζει με σαφήνεια τους ε, περιορισμούς, τα όρια της διαλειτουργικότητας. Είναι κάτι που μάλλον πρόκειται για ένα ζήτημα όπου δεν μπορεί να έχει μόνη αρμοδιότητα ο οργανισμός, αποκλειστική αρμοδιότητα, γιατί εξαρτάται από τη νομική βάση του κάθε πληροφοριακού συστήματος. Κάθε φορά επίσης που εισάγεται ένα καινούριο σύστημα ή μια, μια νέα ευκαιρία επέκτασης της ε, διαλειτουργικότητας, αυτό θα πρέπει να περνάει μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάντοτε πρέπει να έχουν λόγο σε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι σχετικοί περιορισμοί και προδιαγραφέ πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη νομική βάση κάθε ενδεχόμενου νέου τέτοιου πληροφοριακού συστήματο. Γιατί εκεί πρέπει να, να εμπεριέχονται τα εχέγγυα και οι εγγυήσει ε, τη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Would like to intervene on the comments. Ο εισηγητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια συνάδελφοι και Προεδρία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν παρουσίασα το σχέδιο έκθεσης μου, αυτό το έκανα κατόπιν συνεννοήσεως και συζητήσεως με τους και εισηγητές. Δηλαδή, πολλά τα μελήματα και ανησυχίες, όχι μόνο δικά μου, αλλά και των σχεδόν εισηγητών και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο και αυτά που είπε ο κύριος Σάρμπρεχτ για τη λειτουργικότητα είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ ωραία στην τροπολογία περιθμών 9, όπου προβλέπω να απαγορεύεται ε, οποιαδήποτε διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Συμφωνώ και με, τον κύριο, και με την κυρία Λάτφορτ σε ό,τι αφορά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα τα απαντήσω όλα. Θα τα μελετήσω, θα τα επεξεργαστώ. Επιτρέψτε μου να πω τα εξή τρία-τέσσερα πράγματα. Πρώτον, η τροπολογία 14. Μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μπαίνουμε πολύ σε λεπτομέρειες και στον τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά στο άρθρο 14. Μα έχουμε τους λόγους μας για να το κάνουμε αυτό. Ανησυχούμε βαθύτατα για την ασφάλεια των ε, δικτύων αυτών. Ήδη έχω ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω την απάντηση. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, τα νέα είναι πάρα πολύ ανισχυτικά για το σύστημα αυτό. Παράδειγμα, Στο Κάιρο της Αιγύπτου υπάρχει ένα γραφείο που έχει όλες αυτές τις πληροφορίες και όλο το προσωπικό έχει στην τσέπη του ένα σωρό πληροφορίες και στοιχεία με βασικές διευθύνσεις και πρωτόκολλα διαδικτύου για τη διοίκηση, της διοικήσεις των κρατών μελών. Γιατί με τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό κάνουμε εξωτερική ανάθεση και αυτοί οι άνθρωποι εδρεύουν στο Κάιρο. Ανησυχώ πάρα πολύ ε, για τους όρους ασφαλείας. Ε, τώρα, στην Πρατισλάβα. Εξ όσων γνωρίζω, το κτίριο όπου εδρεύουν αυτές οι υπηρεσίες και εργάζονται είναι σε εκτρή κατάσταση ασφαλείας. και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του ΕΣΕΣΤΑ. Και περιμένω την, απο... την απάντηση συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ε, προτιμούσα να έχουμε ασφαλιστικέ δικλείδε στο νομικό κείμενο. Καταλαβαίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει να μην μπουν στο νομικό κείμενο. Ναι, αλλά εδώ ανταπαντώ ότι στο νομοθέτη εναπόκειται να αποφασίσει, ξέρετε, τι θα μπει στο νομικό κείμενο. Εάν θέλει να μπει στι λεπτομέρειε, θα πρέπει να γραφεί και αυτό στι λεπτομέρειε. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Ο νομοθέτη που είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίζει τι θα γραφεί στο νόμο. Αν έχουμε ανησυχίες και εύλογους φόβους για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορα πράγματα, θα πρέπει να υπάρξουν νομικές διατάξεις για να αποφύγουμε και άλλα προβλήματα στο μέλλον. Δεύτερον, πρόσβαση στα έγγραφα. Μιλώ για τις παραγράφους ε, τροπολογίες 36 και 37. Και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να παραχωρούμε την πρόσβαση στα έγγραφα σε ένα σύστημα, εάν ένα κράτος μέλος δεν συμμετέχει στο σύστημα αυτό. Ξέρω ότι Υπάρχουν και τα λεγόμενα οριζόντια ή εγκάρσια έγγραφα, δηλαδή αφορούν όλο τον κόσμο. Τη διαχείριση του οργανισμού, αυτού καθ' αυτού. Δεν μπορούμε να τα ταξινομήσουμε κάθετα και να τα διαχωρίσουμε. Εντάξει, αλλά σίγουρα και οπωσδήποτε υπάρχουν ε, έγγραφα για κάθε σύστημα ξεχωριστά. Και νομίζω ότι σε αυτή την πρόσβαση θα πρέπει να είμαστε περιοριστική. Μόνο τα κράτη που συμμετέχουν στο κάθε σύστημα. Για τις συμβουλευτικές ομάδες τώρα, advisory groups, προβλέπονται για τα νέα όμως συστήματα επικοινωνιών. Δηλαδή, αν μου λένε ότι τα νέα συστήματα θα πρέπει να μπαίνουν στον οργανισμό με τα νομικά μέσα, όταν θα εγκρίνουμε κάθε φορά το νομικό μέσο, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το εκάστοτε πρόβλημα της συμβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, αν φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό PNR, λίστα προσωπικών δεδομένων ας πούμε, των επιβατών, τέτοιο στυλ, και έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δικαιοδοσία να τα ε, ε, ελέγχει, όταν θα το αποφασίσουμε, τότε θα προσθέσουμε και την αντίστοιχη συμβουλευτική ομάδα, οι ομάδες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε και τελειώνω Είμαι πρόθυμο να συνεργαστώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για άλλες ε, λεπτομέρειε Ό,τι άλλο θέλουν να συζητήσουμε, είμαι στη διάθεσή τους για περαιτέρω διευκρινήσει και άλλα θέματα. Πολλά είναι ακόμα. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Πάντως, και για το διευθυντή πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να ζητήσουμε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουμε. Και τα προβλήματα είναι ότι χρειαζόμαστε agency, ευρωπαϊκό οργανισμό, για να διαχειρίζεται αυτέ τι τράπεζε δεδομένων. Με καλό επίπεδο προστασία δεδομένων, με καλό επίπεδο αποτελεσματικότητα, με καλό επίπεδο ποιότητα ε, στοιχείων που συλλέγονται και οικονομική ε, διαχείριση σχέση κόστος-οφέλειας και όλα αυτά. Ελπίζω να ψηφίσουμε όσο γίνεται καλύτερη νομοθεσία για να ε, βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και πάλι ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε την πρόταση αυτή, γιατί αυτό είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και το θέμα αυτό. Ο εισηγητή μίλησε ήδη για το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 12 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ερχόμαστε τώρα στα δύο τελευταία σημεία για το πρωινό, που είναι μια κοινή συζήτηση για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια παραμονής. Και η συγκίτρια και για τις διεκθέσεις είναι η κυρία Ναταλή Κρισβέκ. Α, πρέπει να σας δώσω σύντομα κάποιες λεπτομέρειες. Η απόφαση λήφθη το Σεπτέμβριο του 2008, διαπραγματεύσει έγινε το 2009 και το Νοέμβριο του 2009 μονογράφησαν δύο συμφωνίες. Το Συμβούλιο επέγραψε τη συμφωνία για τη θεώρηση στις 16 Ιουνίου και για την επανεισδοχή δεν μπορεί ακόμα να υπογραφεί η συμφωνία γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ε, τρίμηνη προθεσμία για να προσυπογράψουν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει στην Επιτροπή μας το περιεχόμενο των δύο συμφωνιών. Στη συνέχεια θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας, αν θέλει, να λάβει το λόγο και θα ακολουθήσει συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρώτη το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε και εσείς η ίδια το σήμα για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες αυτές δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την ε, συνεδρίασή του της 1ης Σεπτεμβρίου του 2008 Πράγμα που ήρθε πράγμα που προέκυψε αμέσως μετά τη σοβαρή κρίση, την ανάμνηση της οποίας διατηρούμε όλοι στο μυαλό μας. Προφανώς οι ηγέτες των κρατών και των κυβερνήσεων ήθελαν να δώσουν στον λαό της ήθελαν να στείλουν στο λαό της Γεωργίας έντονο δείγμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, συγκεκριμένα μεταξύ πολλών άλλων πρωτοβολιών ε, που ανελήφθησαν εκείνη την εποχή ε, στον τομέα της διευκόλυνσης της κινητικότητας των ατόμων και των διαπροσωπικών επαφών. Για το λόγο αυτό μας ζητήθηκε τότε να ξεκινήσουμε αυτές τις αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που όπως είπε και η ίδια η Πρόεδρος ήταν σχετικά σύντομες, γιατί αφού τον Οκτώβριο του 2008 το Συμβούλιο είχε δώσει την άδειά του να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές, χρειαστήκαμε λιγότερο από ένα χρόνο για να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου με τους εταίρους μας από την Γεωργία. Οι συμφωνίες, είτε αυτή που αφορά την απλούστευση, είτε αυτή που αφορά την επανεισδοχή, είναι και οι δύο αρκετά κοντά ε, στο κλασικό πρότυπο των τέτοιων συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσο αφορά τη συμφωνία διευκόλυνσης ε, της έκδοσης θεωρήσεων Schengen, η διαδικασία αυτή θα προσφέρει στους υπηκόους της γεωργίας θα τους διευκολύνει, όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης, παρέχεται μια μέγιστη προθεσμία για την έκδοση της σχετικής θεώρησης, 10 ημέρες, στη μειωμένη τιμή των 35 ε, με 60 ευρώ ή και δωρεάν ακόμα για ορισμένες κατηγορίες ε, ταξιδιωτών, ε, δημοσιογράφοι, φοιτητές, άτομα που συμμετέχουν σε πολιτισμικές, καλλιτεχνικές, ή επιστημονικές διοργανώσεις ε, για τα παιδιά των συνταξιούχων ή για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Οι ίδιες κατηγορίες ε, επιβατών, ταξιδιωτών θα ε, απολαμβάνουν κι άλλων διευκολύνσεων, πάντοτε στο πλαίσιο της απλούστευσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ε, βίζας ή ακόμα και έκδοση θεωρήσεων ε, με πολλαπλούς αποδέκτες. Ο υπολογιζόμενος αντίκτυπος της συμφωνίας με βάση τα αιτήματα για έκδοση θεωρήσεων που καταγράφονται είναι 60.000 ταξιδιώτες ετησίως. 60.000 πολίτες της Γεωργίας ετησίως ζητούν την έκδοση μιας θεώρησης Schengen για να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν τον χώρο Schengen. Προσφέροντας λοιπόν αυτήν την διευκόλυνση στην κινητικότητα των ταξιδιωτών, ο αριθμός τους μπορεί και να αυξηθεί στο μέλλον. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις φυσικά, η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση της υποχρέωσης ε, ε, θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, πράγμα που θα διευκολύνει και τις επίσημες επαφές μεταξύ των γεωργιαγωνών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Κυρία Πρόεδρε, ενδιαφέρον είναι ότι μετά από την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας αυτή η διευκόλυνση στην ε, διαδικασία έκδοσης των θεωρήσεων είναι η πρώτη, θα είναι η πρώτη, όπου το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Σίγουρα μια πολύ καλοδεχούμενη θεσμική εξέλιξη. Όπως πάντοτε στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής που αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή, αυτές οι συμφωνίες διευκόλυνσης πάει μαζί, συνοδεύεται με μια συμφωνία επανεισδοχής. Και εκεί ε, ακολουθείται το κλασικό μοντέλο, το το οποίο είναι πολύ κοντά στις συμφωνίες επανεισδοχής που έχουμε διαπραγματευτεί και συνάψει με έναν αριθμό τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται μια τέτοια συμφωνία όχι μόνο στους υπηκόους της Γεωργίας ε, που διαμένουν παράνομα, αλλά και σε κάθε υπήκο τρίτου, τρίτης χώρας για τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι διήλθε με βεβαιότητα μέσω της γεωργίας πριν να, πριν να εντοπιστεί όσο διαμένων παράνομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας επιτρέπουν να μετρήσουμε το, τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ανάγονται στο 2007 και μιλούν για 4.800 υπηκόους της Γεωργίας οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο εντοπίστηκαν ως διαμένοντες παράνομα στην επικράτεια κάποιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και που μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής, γιατί είναι η δεύτερη τέτοια συμφωνία. Υπήρξε μια παρόμοια ε, συμφωνία όπου ζητήθηκε και η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για το Πακιστάν ε, τότε το Κοινοβούλιο μας είχε ζητήσει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της ε, προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας και επίσης προσοχή να δώσουμε στο σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κείμενα, τα ισχύοντα στον τομέα του διεθνούς δικαίου Όπως θα θυμάστε, η Ευρωπαϊκή, η Γεωργία είναι, έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης του 1950 ε, του 1951 για τους πρόσφυγες. Ε, την υπέγραψε νομίζω το 1990. Πιστεύω ότι οι συμφωνίες αυτές θα τύχουν πολύ ευνοϊκής ε, υποδοχής από την κυβέρνηση και ιδίως από το λαό της Γεωργίας. Θα το εκλάβουν αυτό σε ένα απτός δείγμα αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι θα υπάρξει υποστήριξη για τις συμφωνίες αυτές και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα μας μιλήσει και η Προεδρία γι' αυτό σε λίγο. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Λεπρόεδρος, και τώρα δώσουμε το λόγο στην Ισπανική Προεδρία. Ε, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα να πούμε κάτι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τη συμφωνία. Όπως ε, εξήγηκε το περιεχόμενό της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντελεχώ, εμείς Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το επιδευθέν αποτέλεσμα κατόπιν των ε, δραματεύσεων, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να ε, συμφωνηθεί αυτή η επανεισδοχή κάποια χώρα. Το δούλεψε πάρα πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετικά σύντομα να μας πει κατά πόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτής της συνένεσης, ώστε να ακολουθήσουμε αυτό το κλασικό μοντέλο της επανεισδοχής. Αναβάνουν όλοι τις ε, ευθύνε τους και επίσης θα πρέπει να τηρηθεί η σύμβαση της Γενέβης και οι άλλες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς όπως παραμένουν σε αυτές οι η ε, διατάξη της συμφωνίας και γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Απλώς θέλουμε να σας πούμε ότι, στο είπε το Συμβούλιο ε, για την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά αυτή την ρήτρα για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι όπω γνωρίζετε, σύμφωνα με τι συνθήκε, ε, τα όσα περιχόνται είναι παραδείγματα η Ιρλανδία έχει τρει ε, μήνε, τόσο ώστε να πει κατά πόσον θέλει ή όχι να συμμετάσχει για αυτέ τι ρυθμίσει για την μετανάστευση. Εξέπνευσε η συνθήκη και πρέπει να μάθουμε αν θα πούν ναι ή όχι. Επίση, έχουμε από την άλλη μεριά τα των θεωρήσεων διαβατηρίου όπου συμμετέχουν αυτέ οι δύο χώρε. Οπότε είναι δυνατόν εκεί να κάνουμε επίσημη κίνηση. Πάντω, σα ξαναλέω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο τη συμφωνία. Και θα ήταν καλό να δώσει το πράσινο φω και το κοινοβούλιο τώρα όσον αφορά αυτή τη συμφωνία για τη διευκόλυνση χορηγή θεωρήσεων. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να δώσετε τη σκητάλη στον συνάδελφο ο οποίος χειρίζεται ε, το συγκεκριμένο θέμα για την Προεδρία. Ε, ε, δεν έχω να προσθέσω παρά μόνο πολύ λίγα σχετικά. Θα μπορούσα ίσως να πω ότι παρόλο που δεν είναι αμυγός θέμα θεωρήσεων, την 1η Σεπτεμβρίου του 2008 το Συμβούλιο αποφάσισε και την ενίσχυση των σχέσεων με τη Γεωργία και τη σύναψη συμφωνία για ένα χώρο ε, ελευθέρων συναλλαγών με ένα κεφάλαιο συμφωνίας ε, σύνδεσης που θα αρχίσει η διαπραγμάτευση γι' αυτό το πιθανότερο του φέτος τον Ιούλιο. Μαζί με άλλες δύο χώρες, με τις ε, ε, ε, χώρες του Νοτιού Καυκάσου, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν. Παρόλο που το Αζερβαϊτζάν δεν είναι μέλος του ΠΟΕ ακόμα και δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί συμφωνία τέτοιου τύπου ελευθέρων συναλλαγών. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και ερχόμαστε τώρα στα μέλη της Επιτροπής. Η συγγήτρια πρώτα βεβαίως, η κυρία Γκρισμπέκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για αυτές τις δύο συμφωνίες. είναι ταυτόχρονα μια παρουσίαση του θέματος αλλά και η λήξη του θέματος. Γιατί παρόλο που μπορούμε να συζητήσουμε λίγο τις ε, διατυπώσεις, ε, δεν έχω τίποτα να πω για τις ε, τεχνικές προδιαγραφές αυτών των δύο συμφωνιών. Μόνο διανύουμε ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Ε, νομίζω ότι ζούμε μια ιστορική πρόοδο αυτή τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα και μια κοινωνική, πολιτική, θεσμική, τεχνική πρόοδο. Ποια είναι, ε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την θέση του Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια πολύ σαφής βούληση προσέγγισης της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκφράζεται μέσα από μια σειρά σημαντικών πολιτικών ε, πρωτοβουλειών, τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου, στις εταιρικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το σημαντικό τραυματικό επεισόδιο για τους Γεωργιανούς αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το συμβάν, η εισβολή της Ρωσίας στην Νότια Οσετία το 2008, αυτή η εισβολή λοιπόν έπληξε, μάλλον έθιξε την πολιτική γυτνίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαίνοντα τρόπο, αλλά πάντως πάρα πολύ σύντομα ε, ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόκληση αυτή και από το φθινόπωρο του 2008 μετά και την έγκριση του Συμβουλίου και την θετική γνώμη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινήσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Τα ευρωπαϊκά όργανα εξέφρασαν τις θέσεις τους. Ε, θυμάμαι την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος ε, για τον Νότιο Κάυκασο. Ε, ζητήσαμε μια ενεργό δραστηριοποίηση στην γεωγραφική αυτή περιοχή για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή Μια σειρά λοιπόν κινήσεων που δείχνουν τη διαδικασία προσέγγισης ε, ως αποτέλεσμα της οποίας η γεωργία στρέφεται περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά προς άλλους ε, παράγοντες της διεθνούς κοινής. Ε, οι δύο συμφωνίες ταυτόχρονα ε, εγκρίνονται, αν και νομίζω ότι η Συμφωνία Επανεισδοχής θα προηγηθεί τεχνικά της Συμφωνίας Απλούστευσης της Έκδοσης ε, Θεωρήσεων. Μιλήσαμε για τις κατηγορίες των δικαιούχων. Με μεγάλη σαφήνεια περιγράφονται όλα αυτά στις δύο συμφωνίες. Λοιπόν, εκ προημίου θα διευκολυνθεί αυτή η συνεργασία. Ο αριθμός των προσώπων δεν είναι και τόσο σημαντικός που διακινείται. Σίγουρα όμως μετά από την έγκριση αυτών των δύο συμφωνιών θα αυξηθεί. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την περαιτέρω εδραίωση των σχέσεών μας με τη Γεωργία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τη γεωργία μέσω των και άλλων διαπραγματεύσεων και άλλων συμφωνιών. Πάντως έχουμε εδώ μια πρώτη ε, περίπτωση όπου θα δοθεί σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου μετά την ε, μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ναι, υπάρχουν ε, στοιχεία ε, σύγκρισης ενδεχομένως με το Πακιστάν, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Ε, η Γεωργία έχει υπογράψει όχι μόνο τη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό θα σημάνει την αρχή, σημα, σημαίνει την αρχή αυτού που αποκαλέσαμε ως ε, κλασικό μοντέλο συμφωνίας. Ε, είναι οι πρώτες συμφωνίες που θα ακολουθήσουν αυτό το κλασικό μοντέλο ε, για τις συνθήκες ασφάλειας, τις νόμιμες προϋποθέσεις και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μας θα συμφωνήσει. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ντανοκα που έχει ζητήσει να πάρει το λόγο. Yes. Is it Ευχαριστώ. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μου υποστηρίζει πάντα τα βήματα διευκόλυνσης, απελευθέρωσης, δηλαδή ε, της ε, χωρίς θεωρήσεων ευατηρίων με τους εταίρους μας. Είναι κλασική η μορφή αυτής της συμφωνίας, αλλά είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την επανιστογή και τις, συνθήκες, και τις συμφωνίες επανεισδοχής. Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστά κατάλαβα αυτό που είπατε. ότι είναι περίπου 5.000 εκείνοι που καλύπτονται από τη συμφωνία αυτή επανεισογής και ζουν σήμερα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε για την σωματική τους ακεραιότητα, αν ε, επαναπροωθηθούν, εν πάση περιπτώσει, ή εκδοθούν ή απελαθούν προς τη Γεωργία. διότι ξέρουμε ότι ε, στα διάφορα καθεστώτα ε, στα διάφορα, μάλλον σε, διάφορα κράτη έχουν διαφορετικό καθεστώς οι άνθρωποι αυτοί, διαφορετικά διαφατήρια. Ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, απειλείται η ζωή τους. όταν θα επιστρέψω στη χώρα της. Ο κύριος Μπούσουτιλ. Ευχαριστώ η συνάδελφός μου Μόνικα Μακοβέη είναι σκιώδη συγγήτρια για τις δύο αυτές εκθέσεις και απουσία της ε, θα ήθελα να λάβω το λόγο. Η θέση μου διαφέρει λίγο από τις προλαλήσεις εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τις δύο συμφωνίες. Είναι πολύ καλή στρατηγική όταν ε, συνοδεύονται οι ε, συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης ε, θεώρησης με συμφωνίες επανεισδοχής. Γιατί η μία συμφωνία ενισχύει την αξιοπιστία της άλλης. Και επίσης είναι πολύ καλή στρατηγική να συνεχίσουμε αυτές τις συμφωνίες για την επανεισδοχή, γιατί αυτό έρχεται να υπογραμμίσει τη σημασία της κοινή πολιτικής που ακολουθούμε για τη μετανάστευση. Και σήμερα το πρωί αρμόδια υφυπουργός ε, της Ισπανικής Προεδρία το είπε. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση της πολιτικής μας για τη σωστή, την νόμιμη μετανάστευση με την πολιτική για τη λάθρο μετανάστευση. Είναι δύο σκέλη της πολιτικής μετανάστευσης και αν δεν επικρατεί η ισορροπία τότε δεν θα έχουμε καμία αποτρεπτική ισχύ και θα είναι κίνητρο να έρχεται ο κόσμος παράνομα και να παραμένει παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και σε διεθνή συνεργασία είναι κρίσιμο να συνεργαζόμαστε με τα κράτη αυτά τα τρίτα και για την ε, αξιοπιστία και για την ισχύ των συμφωνιών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ασφαλιστικές δικλείδες, όπως ε, μόλις είπε η συγγήτρια, το γεγονός ότι η Γεωργία εδώ ε, είναι συμβαλόμενο μέρος ε, των σημαντικών συμβάσεων της ΕΝΕΒΙΣ και της ΕΣΔΑ, ε, θα πρέπει να μας καθησυχάσει ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και χέγγια και δεν ε, απειλείται η σωματική ακαιρεότητα των ε, προσώπων που επαναπροωθούνται. Κύριε Πρόεδρε, συνιστώ υπερψήφιση εξ ονόματος της ομάδας μου. Ευχαριστώ Σάιμον. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στην ερώτηση που της έγινε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους παρεμβαίνοντες για την ε, γενικότερη υποστήριξη προς το διάβημα της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει. Μερικά, μερικές διευκρινήσεις για, το, τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Τζούνκα. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω αυτό που είπα γενικά για τις συμφωνίες της επανεισδοχής, για το τι είναι, ιδίως στο πλαίσιο της συζήτησης, στο πλαίσιο της, συζήτησης της συμφωνίας με το Πακιστάν. Η συμφωνία επανεισδοχής είναι μια διαδικαστική συμφωνία, η οποία οργανώνει τη διαδικασία και τη διευκολύνει τη, την ε, διαδικασία επαναπατρισμού υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που λαμβάνεται απόφαση απομάκρυνσης του ενδιαφερόμενου, απόφαση η οποία λαμβάνεται από κάποιο κράτο μέλος. Η απόφαση αυτή απομάκρυνσης πλαισιώνεται και θα πλαισιώνεται από την οδηγία για την επιστροφή, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους και που είναι καρπός ε, κοινή εργασίας των συνομοθετικών οργάνων, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Λοιπόν, όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μια απόφαση να απομακρύνει ένα συγκεκριμένο άτομο, γενικά και σύμφωνα με τη συμφωνία, ε, υποχρεώται να εφαρμόσει, δεσμεύεται από όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και από όλους τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου. Υπάρχουν, υπάρχουν τα δίκαια αυτά και εφαρμόζονται στη διαδικασία επανεισδοχής. Δεν πλήττονται τα δικαιώματα αυτά, δεν περιορίζονται. Τώρα, ειδικά για τη γεωργία, επιβεβαιώνω τον αριθμό που είπατε, τον ίδιο περίπου αριθμό ανέφερα και εγώ, είναι μια εκτίμηση. Δεν είναι εκτίμηση, είναι στατιστικά στοιχεία που βασίζονται το 2007 ε, και αφοράν, αφορούν τα στατιστικά αυτά στοιχεία τον αριθμό των παράνομα διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, 4.800. Οι άνθρωποι αυτοί, εάν ίσχυε τότε η Συμφωνία Επανεισδοχής, θα είχαν επαναπατριστεί εφαρμόζοντας όλες τις εγγύησεις της Συμφωνίας και θα ίσχυαν στη Γεωργία όλες οι εγγυήσεις τις οποίες έχει προσυπογράψει η Γεωργία βάσει των διεθνών συνθήκων που έχει ε, υπογράψει, τη Σύμβαση της Γενέβης ε, για τους πρόσφυγες, τη Σύμβαση για την ανθρωπιστική μεταχείριση, τη Σύμβαση για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επομένως, ε, έτσι μπορούν να καθησυχαστούν και οι ηγέτες των κρατών μελών όταν λαμβάνουν την απόφαση απομάκρυνσης, ε, ε, αλλά διασφαλίζονται και καθησυχάζονται και οι αρχές της γεωργίας όταν θα υποδεχθούν πίσω ε, το... τα εν λόγω άτομα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα, ζητήσω την... θα ρωτήσω την εισηγήτρια. Θέλετε να απαντήσετε? Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις αυτές τις σαφείς απαντήσεις σας που όλα αυτά νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται για αυτή τη συμφωνία για να μπορέσουμε με αυτό το διεθνές κείμενο όσον αφορά τη γεωργία να κάνουμε ό,τι μπορούμε και έτσι να παρασχεθούν κάποιες εγγυήσεις για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, οδηγία αυτή για την επανεισδοχή. Βέβαια δεν είναι και πολλοί συνάδελφοι εδώ, περιμένω τη δική τους επιστροφή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, ίσως φαντάζομαι το φθινόπωρο να βάλουν τελευταίες πινελιές σε αυτή τη διαδικασία και, και τις δύο συμφωνίες οι οποίες πάνε χέρι-χέρι. Επομένως το σχέδιο του κειμένου σας πρόκειται μετά να παρουσιαστεί μετά το καλοκαίρι. Τώρα επομένως κύριε Σωτήρη, λήξη της συνεδρίασης και θα συνεχίσουμε στις 4.30. Αφού γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια.